Okay, colleagues, Αγαπητοί συναδελφοί, ας ξεκινήσουμε. Έχετε την ημερήσια διάταξη, εγκρίνετε. Αν δεν έχετε να προτείνετε καμιά αλλαγή, διαφορά, τίποτα. Έχουμε να εγκρίνουμε τώρα τα πρακτικά τη 8η Μαρτίου 2010, 22η-23η Μαρτίου 2010 και 26η-27η Απριλίου 2010. Σχόλια για τα πρακτικά. Αν έχετε τώρα. Όχι από ό,τι βλέπω. Καλώς. Μία ανακοίνωση έχω να κάνω. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι τον Ιούνιο στο Στρασβούργο 7 με 8.30 θα έχουμε έκτακτη συνεδρίαση για να ψηφίσουμε εκθέσεις. Σας υπενθυμίζω ότι και 21 Ιουνίου θα συνεδριάσουμε. 3 το απόγευμα και την επόμενη μέρα πρωί και απόγευμα. Αυτές είναι οι ανακοινώσεις που έχω να κάνω. Περνάμε λοιπόν στα θέματα που θα εξετάσουμε σήμερα. Το σημείο 4 είναι η έκθεση του κυρίου Hans Peter Μάρτιν για την διασύνδεση των μητρών επιχειρήσεων. Πολύ ενδιαφέρον. Οπότε, παρακαλώ τον εισηγητή να μας παρουσιάσει το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Είναι πιο ενδιαφέρον το θέμα από ό,τι νομίζετε, κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Είχαμε μία συζήτηση για να ολοκληρώσουμε, για να, κάνουμε το, για να γίνει ο φάκελος αυτός πολύ πιο αποτελεσματικό και να προχωρήσουμε ταχύτερα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα του συναδέλφου οι οποίοι υπέβαλαν τροπολογίες. Äh, και ενσωμάτωσα τις ε, τροπολογίες ε, που αναφέρθηκαν στη συζήτηση ιδιαίτερα του συναδέλφου κυρίου Μπούλμαν και προσπάθησα να ανταποκριθώ στα αιτήματα των συναδέλφων. Έχω δύο προβληματάκια. Το ένα είναι η τροπολογία 4 του συναδέλφου Πίτερ Ζήμον που προτείνει, που επιμένει όλοι μέσα από το δίκτυο να λάβουν πληροφορίες ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα γίνει αυτό λοιπόν, δεδομένου ότι εμείς θέλουμε ένα κοινά προσβάσιμο δίκτυο, ένα κοινά προσβάσιμο μητρό, αλλά εάν ακολουθήσουμε την πρότασή τους θα χρειαστεί να υιοθετήσουμε ένα, μια επιπλέον διαδικασία Δηλαδή θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και η πηγή της πληροφορίας και πιστεύω ότι αυτό θα είναι υπερβολικά γραφειοκρατικό συν θα δημιουργήσει επιπλέον γραφειοκρατικό άχθος και γι' αυτό ε, ελπίζω αν δεν αποσυρθεί, ως εισηγητής προτείνω να καταψηφίσουμε αυτή την τροπολογία του κυρίου Πίτερ Σίμον δεν, είναι, δεν μπορεί να εφαρμοστεί και θα μας επιβαρύνει με κόστος. Το δεύτερο πρόβλημα που έχω είναι, η τροπολογία η δικιά μου, πέντε. Είχα την άποψη ότι υπάρχει μία σαφής ε, πλειοψηφία επί της ουσίας εδώ στην Επιτροπή, όπως το έχει διατυπώσει πολύ ωραία και ο συνάδελφος Μπούλμαν. Δηλαδή ότι όλοι επισημούμε να βρούμε μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή λύση για αυτό το μητρό το οποίο, η οποία θα είναι ευκολόχρηστη, σαφής ε, και δεσμευτική. <clears throat> Ε, η ομάδα Ευρωπαίων Συντηρητικών δεν θέλουν να δεσμευτούν ως προς ε, την ουσία ε, αυτής της ε, παραγράφου και γι' αυτό θα ήθελα αυτή την τροπολογία να την ψηφίσουμε ξεχωριστά σε δύο τμήματα. Το ένα να είναι το δεσμευτικό και το υπόλοιπο με ξεχωριστή ψηφοφορία. Έτσι ώστε ακόμα και αν ε, δεχθούμε το, την υποχρεωτική φύση ε, να μην ε, τύχει της πλειοψηφίας στην Επιτροπή. Γιατί εν μέρη καλύπτεται και από την τροπολογία του κυρίου ε, Σίμων. Αυτά είχα να παρατηρήσω στις τροπολογίες 4 και 5. Ευχαριστώ για τη, το, τη γραμματεία για τη συνεργασία της και την πολύ επικοδομητική σύμπραξη και προσβλέπω με ιδιαίτερη ευχαρίστηση στην ψηφοφορία. Ευχαριστούμε πολύ. Σχόλια. Μήπω από τους συναδέρφους, ο κύριο Σάιμον, από τους σοσιαλιστέ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον κύριο Μάρτιν για το πολύ χρήσιμο, την πολύ χρήσιμη του σύμπραξη και το υπόβαθρο. Ε, το, το, το, η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει ε, αυτό το μητρό να είναι εμπλουτισμένο επαρκώς, ε, διότι ο στόχος είναι να, να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της πραγματικότητα στην Ευρώπη. Και γι' αυτό διαφορετικά από τον συνάδελφο, κύριο Μάρτιν, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ένα σημείο επισκόπησης όπου μπορούμε να εξασφαλίσουμε την πιστότητα των στοιχείων, εξακριβώνουμε δηλαδή κατά πόσον τα στοιχεία αυτά είναι αληθή, διότι διαφορετικά θα δοθεί η εντύπωση στον κόσμο ότι δεν υπάρχει ουσία στο μητρό αυτό και είναι απλώς εικονικό. Ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι εάν δεν υπάρχει μια τέτοια υποχρέωση επικαιροποίησης των στοιχείων ε, και εξασφάλισης της ακρίβειας, της πιστότητας των στοιχείων. Πρόκειται λοιπόν εδώ για ουσιαστική ερώτηση. Δηλαδή, θέλω να δημιουργήσω ένα μέσο το οποίο θα μας προσφέρει μια πάρα πολύ σωστή και πιστή εικόνα όλων των επιχειρήσεων στην Ευρώπη ή δεν το θέλω αυτό. Εάν δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ε, πιστότητα και την ακρίβεια των στοιχείων που θα περιέχει αυτό το μητρό, είναι το νόημα. Ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή, τον κύριο Hans Peter Μάρτιν, για την έκθεσή του. Αλλά θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό που είπε ο κύριο Σίμων. Θέτει ένα θέμα αρχής. Οι κόστους Αναρωτιέμαι. Από πλευράς του ΕΛΚ συμφωνούμε επί της αρχής ότι ένα τέτοιο λειτουργικό μητρό είναι πολύ καλό για τις επιχειρήσεις. Όμως μεταξύ των χωρών μελών υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα. Στη χώρα μου, τη Λετωνία για παράδειγμα, που είμαστε καινούργοι, ξεκινήσαμε από το μηδέν πριν από 20 χρόνια και έχουμε ένα αρκετά μετριόφρον τέλο πάντων σύστημα διασύνδεσης μητρών επιχειρήσεων. Όλες οι χώρες μέλη δεν έχουν ε, εξίσου ε, προχωρημένα επίπεδα διασύνδεσης μητρών, ορισμένοι πολύ πιο πρόσφατα ξεκίνησαν. Οπότε, εμείς λέμε από το ΕΛΚ ότι αν γίνει υποχρεωτικό, δεσμευτικό αυτό, ποιος θα πληρώσει, πώς θα πληρωθεί. Συμφωνούμε λοιπόν επί του πνεύματος, επί της αρχής της πρότασης, αλλά το ΕΛΚ δεν θα στηρίξει τον υποχρεωτικό χαρακτήρα ενός τέτοιου μητρώου. Οπότε γι' αυτό θέλω να ξέρω το κόστος ποιο θα είναι στα κράτη-μέλη, για να δούμε και το Συμβούλιο δηλαδή τι θα πει. Εμεί πιστεύουμε ότι δεν θα συμφωνήσει το Συμβούλιο να πληρώσουν οι χώρες μέλη. Αυτό πρέπει να δούμε. Ας αφήσουμε λοιπόν το δεσμευτικό στην πάντα προς το παρόν. Ευχαριστούμε. Στρέτσεκ, μέρους των Ευρωπαίων Συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, δεν έχω να προσθέσω πολλά σε αυτά που είπε ο Χάνς Πέτερ Μάρτιν. Εκεί που διαφέρουμε κάπως όσον αφορά την προσέγγισή μας είναι το εξής. Εμείς πιστεύουμε ότι η διασύνδεση εμπορικών μητρών, μητρών επιχειρήσεων πρέπει να διασφαλίζει ότι το σύστημα μπορούμε να το πληρώσουμε, ότι είναι αποτελεσματικό και θα είναι αποτελεσματικό στο μέλλον και ότι βασίζεται σε όσο γίνεται λιγότερη γραφειοκρατία. Αυτό έχει να κάνει και με το κόστος βέβαια. Κόστος το οποίο πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο χαμηλό. Και εφόσον γνωρίζουμε ότι διαφορετικά κράτη-μέλη έχουν διαφορετικά συστήματα, δεν μπορούμε να δεχτούμε μια τόσο απαιτητική πρόταση. Γι' αυτό και λέμε ότι ίσως το Συμβούλιο βρει μια καλύτερη διατύπωση. Εμείς πάντως, από τη δικιά μας την πλευρά, θέλουμε περισσότερη ελευθερία, περισσότερο περιθώριο ελιγμών στις χώρες μέλη. Και σίγουρα θα συμφωνήσει και το Συμβούλιο με αυτό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπόμεν έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε εισηγητή. Με την εργασία του συναδέλφου Πίτερ Ζήμων είναι σαφές ότι η ομάδα μας προσεγγίζει το θέμα αυτό με μεγάλη σοβαρότητα. Δεν είναι δευτερεύον θέμα, διότι πιστεύουμε ότι ένα σωστό μητρό επιχειρήσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εσωτερικής αγοράς. Γιατί, διότι όλο και περισσότερη νομοθεσία ε, δημιουργείται και μπορούμε να την υλοποιήσουμε ικανοποιητικά όταν ε, γνωρίζουμε ακριβώς ε, ποιος κάνει τι και δει στο διασυνοριακό πεδίο. Σας θυμίζω το μεγάλο τομέα των υπηρεσιών η οδηγία των υπηρεσιών από την προηγούμενη θητεία δεν μπορεί να εφαρμοστεί εάν δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι, ποια είναι η δέσμη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που άπτεται αυτού του θέματος Ποια νομοθεσία είναι καθαρά εθνική, ποια μπορεί να εφαρμοστεί διασυνοριακά και Πολλές φορές δεν γνωρίζουμε, δεν μπορεί να εφαρμοστεί η νομοθεσία διότι δεν γνωρίζουμε πού να απευθυνθούμε. Ποια είναι η διεύθυνση της, ε, ε της επιχείρησης, της εμπλεκόμενης επιχείρησης, πού βρίσκεται, πού εδρεύει και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνω ότι η γραφειοκρατία πρέπει να, να μείνει σε χαμηλά επίπεδα, αλλά εάν δεν εφαρμόσουμε κοινά πρότυπα στο μητρό αυτό, ε, τότε ε, θα, δεν θα ε, εφαρμόζονται σωστά και οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς. Όποιος είναι κατά αυτού του μητρό είναι και κατά της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Δεν θέλω αύριο σε αυτό το ουσιαστικό θέμα να δημιουργηθεί μία, να υπερψηφιστεί η έκθεση αυτή τυχαία, έτσι κατά λάθο δηλαδή. Θέλω ενσυνείδητα να υπερψηφίσουμε αυτήν την έκθεση. Ε, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αμφιβολίες, δεν πρέπει να υπάρχουν αμφιβολίες και όσες ε, υπάρχουν δεν τις καταλαβαίνω. Θα ήθελα όσες ομάδες αμφισβητούν ε, την ουσία αυτής της πρότασης να μας εξηγήσουν τη θέση τους για να ξέρουμε πού θα βαδίσουμε αύριο. Ο Σμιτ εκ μέρους του σκιώδησης των σκιωδών εισηγητών. Ναι, ελπίζω κύριε Πρόεδρε. Θα προτιμούσα να ήταν εδώ ίδια, τι να κάνω. Τέλο πάντων, έχω τουλάχιστον εδώ κύριε Μπόμεν τον κατάλογο με την ψηφοφορία. Και έχουμε κάποια προβλήματα με την παράγραφο 4 του αρχικού κειμένου που αναφέρεται στην ομάδα Στόιμπερ. Και στην παράγραφο 5, τροπολογία 5, που υπάρχει έτοιμα για κατατμήματα ψηφοφορία από το ECR. Εμείς καταψηφίζουμε το πρώτο τμήμα και υπερψηφίζουμε το δεύτερο. Και η τροπολογία 6 του Πίτερ Σίμον, νομίζω. Και είναι περίπου συμβατή με την 5. Εδώ μπορεί να ψηφιστεί ως προσθήκη. Αλλά δεν τη διχόμαστε. Εμεί θέλουμε το αρχικό κείμενο. Στα άλλα έχουμε συν. Εντάξει κύριε Μπούμαν, σας ικανοποιεί αυτό. Παρακαλώ κύριε Μπούμαν. Δεν θέλω να προτρέξω του σκιώδη εισηγητή. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο να συζητήσει ο με τους σκιώδη εισηγητής μετά το τέλος της σημερινή συνεδρίασης για να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. Και ε, εν κατακλείδη, ο εισηγητής. Βεβαίως, ευχαριστώ κύριε Πούλμαν, θα το κάνω αυτό. Αλλά και για λόγους δημοσιότητας πιστεύω ότι όλα πρέπει να είναι απόλυτα διαφανή. Ε, δεν σας κατάλαβα πολύ καλά κύριε Σμιτ, γιατί υπάρχει ακόμα σάφια στον κατάλογο ψηφοφοριών. Οι φιλελεύθεροι θέλουν το μητρό αυτό να είναι υποχρεωτικό ή όχι είναι υπέρ της υποχρεωτικής φύσης. Α, υπέρ. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι το ουσιαστικό θέμα. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Ο κύριος Ζήμων, οι σοσιαλδημοκράτες, ε, πράσινοι και φιλελεύθεροι και ο εισηγητής, ε, η πλειοψηφία δηλαδή πιστεύω, είναι υπέρ της υποχρεωτικής φύσης χωρίς να γνωρίζουμε ακόμα ακριβώς πώς θα ελαχιστοποιήσουμε το γραφειοκρατικό κόστος. Παρακαλώ, να, να είσαστε σαφείς. Είμαι υπέρ της υποχρεωτικής φύσης, δεν είμαι κατά του υποχρεωτικού Γι' αυτό θέλω να βρω έναν τρόπο να ανταποκριθώ και στο, στην ανησυχία του κυρίου Ζήμουν για την γραφειοκρατία. Ε, να υποφύγουμε το επιπλέον κόστος. Ελπίζω αύριο να υπερψηφιστεί, διότι βεβαίως εμείς ε, θέλουμε να ε, υπάρχει ένα πρότυπο σε αυτό το, να είναι πρότυπο αυτό το Μητρό. Ελπίζω αύριο, όπως σας είπα, να υπάρξει πολιτική πλειοψηφία και όχι τυχαία να υπερψηφιστεί αυτή η πρόταση, η τροπολογία. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, είμαι ευτυχής που βλέπω ότι υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στις ομάδες και αύριο λοιπόν θα το ψηφίσουμε αυτό το θέμα, αυτή την έκθεση. Περάσουμε στο σημείο 5 τώρα που αφορά την εγγύηση της ανεξάρτητης, ε, τη διασφάλιση μάλλον ανεξάρτητων εκτιμήσεων. Αυτό έχει αναβληθεί λοιπόν. Έχουμε το 6. Έχουμε μια γνωμοδότηση για την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων από τον κύριο Άσλι Φόξ για τη δημογραφική πρόκληση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Έχετε το λόγο κύριε Φόξ. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντα τη Γραμματεία για τη βοήθειά τη στην προετοιμασία αυτή τη ε, ε, γνωμοδότηση. Οι δημογραφικέ αλλαγέ δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο, αλλά οι επιπτώσει τη ε, στη δημόσια οικονομία είναι πρόσφατο, γιατί λόγω τη οικονομική ύφεση είναι ακόμα πιο έντονο το πρόβλημα. Εμεί έχουμε αναλάβει την ευθύνη για να εστιάσουμε στην βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών σε σχέση με τις συνταξιδοτικά συστήματα ώστε να ανταποκριθούμε στη δημογραφική πρόκληση. Όπως με όλες τις νομοδοτήσεις, για να είμαστε αποτελεσματικοί, θα πρέπει να εστιάσουμε στο να δώσουμε στην, στην Επιτροπή Αποσχόληση μια σαφή οικονομική χρειά που εμπίπτει στις δικές μας αρμοδιότητες και θα ήθελα να ζητήσω από τους υπόλοιπους σκιώδεις και του συναδέλφους να το λάβουν αυτό υπόψη όταν θα συντάξουν τις τροπολογίες τους. Είναι σαφές ότι τα φορολογικά συστήματα και τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας είναι θέματα ε, εθνικής αρμοδιότητας. Ρόλος μας είναι, θεωρώ, να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να προβούν στις αρμο... απαραίτητες δράσεις ώστε να διαχειριστούν τις δημογραφικές αλλαγές. Μια γυράσκουσα, ένας γυράσκων πληθυσμός σημαίνει ε, την πρόθεση ε, των προσωπικών, ιδιωτικών μάλλον ασφαλιστικών συμβολέων αλλά και συμβολέων ασφάλισης για σύνταξη καθώς και των ιδιωτικών αποταμιεύσεων θα πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι και πιο, να ανταποκριθούμε στι δημογραφικέ αλλαγέ, να διασφαλίσουμε ότι οι πιο ηλικιωμένοι θα μπορούν να εργαστούν όσο το επιθυμούν εντό τη αγορά εργασία, να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν οικονομικά αντικίνητρα στην δημιουργία μιας οικογένεια. Εδώ θα κλείσω, κυρία Πρόεδρε, και προσβλέπω στη συνεργασία με τους υπόλοιπους σκιώδης για την σύνταξη αυτής της γνωμοδότησης, ώστε να δώσουμε στην Επιτροπή Απασχόλησης μια έκθεση με νόημα. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ που ήσασταν τόσο σύντομος. Να καλέσω τους σκιώδης αν θέλουν να σχολιάσουν. Για το ΕΛΚΑ έχω την κυρία Σάρα Ασέια. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για ένα καλό σχέδιο γνωμοδότησης που περιλαμβάνει πολλές από τους προβληματισμούς που και εγώ ήθελα να αναφέρω για την αλληλεγγύη με τις παλαιότερες γενναίες. Θα πρέπει να προβλέψουμε καλή φροντίδα ε, ώστε να αποφύγουμε το συλλογικό βάρος, υπερβολικό φόρτο στις επόμενες γενναίες επίσης. Καλωσορίζω τη βιωσιμότητα της δημόσιας οικονομίας που είναι μια προϋπόθεση ώστε να μπορέσουμε να μεριμνήσουμε για τους ηλικιωμένου με βιώσιμο τρόπο. Και ως, αναφο... ως, του ΕΛΚ για αυτή τη γνωμοδότηση θα υποβάλω κάποιες ε, τροπολογίες. Νομίζω πως θα είναι σύμφωνες με τις δικές σας απόψεις. Τώρα, πόσο σημαντική θα, σημαντικός είναι ο αντίκτυπος της γύρανσης ε, αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσο θα είναι διαθέσιμος ο των πληθυσμός ως εργατικό δυναμικό και ποιο θα είναι το ποσοστό απασχόλησής τους και ποιο θα είναι ο αριθμός των ε, ωρών εργασίας κατά μέσο όρο. Ε, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τους πιο ηλικιωμένους για την συμμετοχή τους στην ε, αγορά εργασίας Μπορεί αυτό να αντισταθμίσει τις αρνητικές, αλλά μπορούμε να αντισταθμίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της γύρενσης με άλλα μέσα. Καταρχήν θα πρέπει να εμποδίσουμε να προλάβουμε τα προβλήματα υγείας. Αν όλα τα αυξημένα χρόνια ε, βίου είναι υγιή αντί για ασθενή, θα είναι πολύ πιο εύκολο να είναι βιώσιμη η κατάσταση. Επίσης υπάρχουν διάφοροι τρόποι για μείωση του κενού ε, βιωσιμότητας αυξάνοντας την παραγωγικότητα στις ε, υπηρεσίες πρόνοιας. Είναι ένα από τα θέματα κλειδιά για να λυθούν τα σορευόμενα προβλήματα. Έχει αναφερθεί από το Υπουργείο Οικονομίας στην Φιλανδία ότι μια ετήσια αύξηση 0,1% στον τομέα του δημόσιου, τομέα, στην παραγωγή μάλλον του δημόσιου τομέα αντιστοιχεί στο να μειωθεί κατά 1% του ΑΕΠ το κενό της ε, βιωσιμότητας. Άλλα μέτρα θα μπορούσαν να είναι η αύξηση του ορίου συνταξιδότησης, η αύξηση του, της γεννητικότητας και η αύξηση των μεταναστών. Ας πούμε θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την στήριξη για τις νέες οικογένειες για να, παρο, για να παροτρύνουμε στην αύξηση της γεννητικότητας. Φαντάζομαι ο τροπολογίε μου θα είναι σύμφωνε λοιπόν με τις βασικές γραμμές του σχεδίου χρηματοδότηση. Σα ευχαριστώ και εξ ονόματο των Σοσιαλιστών έχω τον κύριο Ρουνιό. Madame la Présidente, chers collègues. Αγαπητοί Πρόεδρε, και κυρίες συνάδελφοι, να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την γνωμοδότησή του και εξασφαλίζει σε ένα σύντομο κείμενο τα βασικά στοιχεία και γι' αυτό και εγώ θα μιλήσω άμεσα για τις, ε, τους βασικούς άξονες. Καταρχήν για τα δημογραφικά προβλήματα, όντως έχουν αντίκτυπο στη δημόσια οικονομία και εφόσον πρέπει να χειριστούμε την δημόσια οικονομία, η έκθεση δεν επιμένει αρκετά στη δυνατότητα που έχουν τα κράτη της Ένωσης να αναζητήσουν αποκτήσουν πόρους και το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε κυρίως να τεθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020 όπου θίγονται τα δημογραφικά θέματα χωρίς όμως να τίθεται και το θέμα των ε, αντίστοιχων μέσων δυστυχώς. Ε, έπειτα, η έκθεση αναφέρει τη δυνατότητα του δημογραφικού προβλήματο μέσω μια καλή πολιτική γεννητικότητα. Συμφωνούμε σε αυτό βέβαια, γιατί αν αυξανόταν ο ε, ενεργό πληθυσμό σε μεγάλο βαθμό, τότε το πρόβλημα μεταξύ ανενεργού και ενεργού πληθυσμού θα μειωνόταν. Αλλά από αυτή την άποψη θα πρέπει φυσικά να αποσπαστούν δημόσιοι πόροι για να βελτιωθεί η πολιτική για τι οικογένειε. Αλλά υπάρχει ένα θέμα που η έκθεση δεν το θίγει, δηλαδή μελλοντική αύξηση του ενεργού πληθυσμού, αν αυτή την επιθυμούμε, είναι το θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής φυσικά, που σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να είναι εξαιρετικά δεσμευτική. Να θυμίσω απλά ότι μια ελεγχόμενη μετανάστευση και τακτική μετανάστευση είναι ταυτόχρονα πηγή του ποσοστού ανάπτυξης της Ένωσης, αλλά και ε, φορολογικός πόρος επιπλέον που τελικά θα οδηγούσε στην ελάφρυνση των συνταξιδοτικών συστημάτων. Υπάρχουν δύο μέτρα σημαντικά τα οποία προτείνει η έκθεση και που θα πρέπει να τα συζητήσουμε σε κάποιο βαθμό. Το πρώτο μέτρο που προτείνεται είναι να ευνοηθούν τα ιδιωτικά συνταξιδοτικά ταμεία εις βάρος των δημόσιων ε, και συνταξιδοτικών συστημάτων και να επιστήσουν την προσοχή στο γεγονός ότι υπάρχει το αντικό, η αντική επίπτωση των συγκοινωνούντων δοχείων που θα συνέβαινε αν κάτι τέτοιο γινόταν στην πραγματικότητα. Γιατί εντάξει, μπορεί όντω να ε, ελαφρυνθούν τα δημόσια ταμεία, αλλά τίθεται ένα επιπλέον πρόβλημα όσον αφορά τα νοικοκυριά από την άλλη πλευρά. Γιατί ε, Αυτά θα έπρεπε να πληρώνουν το ιδιωτικό ταμείο συνταξιοδότησης. Μειώνεται λοιπόν η δικιά τους αγοραστική δύναμη, μειώνεται η ανάπτυξη, μειώνονται τα έσοδα από του φόρους και άρα το δημόσιο, ο δημόσιος τομέας θα ζημιωθεί με τη σειρά του αν χρειαστεί τα ιδιωτικά κοινικοκυριά να δίνουν περισσότερα χρήματα σε ιδιωτικά ασφαλιστικά ταμεία. Τέλος, το μέτρο που προτείνει η έκθεση, το άλλο, είναι να συνεχιστεί ο εργασιακός βίος μετά το συνταξιδοτικό όριο. Αυτό θα σήμαινε ότι απλώς μεταφέρονται, μεταφέρεται το βάρος από τα συνταξιδοτικά ταμεία στα ταμεία ανεργία, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ανεργία. Εκτό και αν ε, γίνονταν τέτοιου είδου πολιτικέ που θα αποκαθιστούσαν την πλήρη απασχόληση στην Ευρώπη. Αλλά η έκθεση δεν μιλά για αυτό το σημαντικό θέμα. Και έχω την εντύπωση πω οι σημερινέ περιοριστικέ πολιτικέ που έχουν ευθετεί στα περισσότερα κράτη-μέλη θα μα καταδικάσουν σε ποσοστά ανεργία εξαιρετικά ε, ισχυρά που θα, που θα αποδυναμώσουν και τα συστήματα ε, των ταμείων ανεργία. Εγώ θα καταθέσω διάφορες τροπολογίες με βάση αυτά που είπα και με τα χαρά θα τις συζητήσω με τον εισηγητή και με τους σκιώδει εισηγητέ. Ευχαριστώ. Very good timing by Mrs. Πολύ καλά με το χρόνο ήρθατε κυρία Φαντενφέλτ ακριβώς στην ώρα εκ μέρους της ομάδας σας εφόσον έχετε σχόλια. Μιλάω για να σας δώσω χρόνο να σκεφτείτε και να είσαστε έτοιμοι. Εντάξει, είσαστε έτοιμοι να ξεκινήσετε. Ναι, ευχαριστώ και συγγνώμη που καθυστέρησα. Αλλά όπως ε, και όλοι εδώ μέσα, τρέχω και εγώ από τη μια συνεδρίαση στην επόμενη. Χαίρομαστε πολύ για την έκθεση γενικά, αλλά θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες. Άκουσα τα τελευταία λόγια του προλαλήσαντα για το κατά πόσο είναι βιώσιμο το συνταξιδιωτικό μας σύστημα. Αν δείτε τις συζητήσεις που γίνονται για το ευρώ, για το σύμφωνο σταθερότητας, μία από, ένα από τα πράγματα που συχνά ξεχνάμε είναι ακριβώς ότι τα κράτη-μέλη έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την βιωσιμότητα των συνταξιδιωτικών του συστημάτων. Πάνω σε αυτό λοιπόν θα υποβάλουμε τροπολογία. Θα υποβάλουμε και τροπολογία για να αντικατασταθεί η παράγραφος 6 που ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να στηρίξουν τις οικογένειες στο πλαίσιο των συστημάτων φορολογίας και παροχών. Εδώ δεν νομίζω ότι τα κράτη-μέλη είναι αυτά που πρέπει να πούνε στις οικογένειες και ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πει στα κράτη-μέλη ποιες οικογένειες να στηρίξουν και ποιες όχι. Ωραία. Ο εισηγητής τώρα, ο κύριος Φόξ, για να σχολιάσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους διάφορους κεώδεις για τα σχολιά τους, τα οποία σημείωσα προσεκτικά. Νομίζω πως ε, ε δεν χρειάζεται να απαντήσω προσωπικά, αλλά τους ευχαριστώ και θα είμαι σε επαφή με τη γραφεία τους από εδώ και μπρος. Σας ευχαριστώ. Υποβολή τροπολογιών 4 Ιουνίου και στις 8 Ιουνίου θα είναι η συζήτηση με ψηφοφορία στην Επιτροπή 13 ε, Σεπτεμβρίου. Θα έχουμε χρόνο δηλαδή για να συζητήσουμε ε, το, τις τροπολογίες. Λοιπόν, επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, το 7, είναι η έκθεση του κυρίου Σιγκλούνα για την υιοθέτηση από την Εστονία από το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2011. Και έτσι θα κάνουμε μια γενική εξέταση γιατί έχουν κατατεθεί και τροπολογίες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα θυμόσαστε ότι στην τελευταία συζήτηση που είχαμε εδώ οι περισσότεροι ευρωβουλευτές ε, μας στήριξαν, στήριξαν και την Εστονία για την πολιτική βούληξη, βούληση που επιδεικνύει και για την επιθυμία της να έχει το ευρώ από το 2011. Εννοείται ότι τίθενται κάποια ζητήματα. Το θέμα των στατιστικών είναι αξιόπιστα. Επίσης το θέμα ε, της απασχόλησης. Θέλω να ευχαριστήσω και τους σκιώδεις εισηγητές και τη γραμματεία που συνεργάστηκαν ε, μαζί μου για να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία όσον αφορά τις τροπολογίες. Είχαμε 13 τροπολογίες, 8 από τη Μάρτα Αντρίεσεν, 3 από τον κύριο Κλίντς και 2 από τον κύριο Μίτσελ. Όσον αφορά τις πρώτες 8 λοιπόν τροπολογίες, σέβομαι την άποψη της συντάκτριας που υπέβαλε τις τροπολογίες αυτές, αλλά δεν συμφωνώ βέβαια, γιατί η Εστονία δεν σκοπεύει να αναβάλει την είσοδό της στο ευρώ για κανένα λόγο. Αυτό έχω να πω λοιπόν για τις 8 αυτές τροπολογίες που την ίδια άποψη εκφράζουν. Στο ίδιο καταλήγουν. Έρχομαι τώρα στην τροπολογία Κλίντς για ένα πολύ σημαντικό θέμα. για να μην χρησιμοποιείτε το ευρώ από ορισμένου σαν άλοθη για να ανεβάζουν τις τιμές. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί όντως σε Ορισμένες χώρες έγιναν ιδιαίτερα αισθητέ αυξήσεις στις τιμές, άλλε όχι. Πάντως συμφώνησα με τον κύριο Κλίν. και θα το βάλουμε στην παράγραφο 10, γιατί εκεί έχει θέση, όπου ζητάμε από τις εσθονικές αρχές να ετοιμαστούν καλά για την αλλαγή και πριν και μετά την αλλαγή, οπότε εκεί θα το βάλουμε. Τώρα για τον όρο hidden, κρυφές δεν ξέρω. Πώς είναι δυνατόν. Έρχονται από το κράτος, από πίσω. Έρχομαι τώρα στην τροπολογία για την Eurostat. Σε στενή συνεργασία με τη Στατιστική Υπηρεσία. Κατά τις έρευνές μου, εγώ διαπίστωσα ότι έχει γίνει και ότι η Κομισιόν είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη από την ποιότητα των στατιστικών δεδομένων. Οπότε εγώ θα έλεγα να μπει σαν μέρος της αιτιολογικής σκέψης. Να διασφαλίζει δηλαδή η Κομισιόν ότι σε συνεργασία με τη στατιστική μας υπηρεσία έχει επαληθεύσει η Κομισιόν ότι είναι ιδιαίτερα αξιόπιστα τα στατιστικά δεδομένα. Το λέει η έκθεση αυτή. Οπότε να συμπεριληφθεί σαν ε, ενημερωτικό προς ενημέρωσή μας. Για τον κύριο Μίτσελ τώρα όσον αφορά πάλι τα δεδομένα και τα κριτήρια. Μιλάει για ανεξάρτητα δεδομένα. Τώρα δεν ξέρω τι είναι αυτά τα independent data. Εννοείται ότι έχουν ετοιμαστεί ανεξάρτητα. Έπειτα υπάρχει μια άλλη τροπολογία που ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια προσωμείωση στην περίπτωση της Εστονίας, αν και εκεί γίνει κάτι σαν και αυτό που έχουμε αλλού στην Ευρώπη. Και η τελευταία τροπολογία είναι του κύριου Μίτσελ που δεν έχει να κάνει με την Εστονία. Είναι γενική. Ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ε, έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μιλήσει για τα, τα βήματα τα οποία ε, σκέφτονται να αναλάβουν για να διατηρηθεί στο ελάχιστο ο πληθωρισμός που είναι συνέπεια των χαμηλών επιτοκιών. Λοιπόν, Συμφωνώ με τις τελευταίες τροπολογίες λοιπόν. Απλώς θα βρούμε πριν από αύριο που ακριβώς θα τις τοποθετήσουμε. Ωραία, η Σκιώδης τώρα λέει πρόεδρος, ο κύριος Μίτσελ. Μέρος του παρακαλώ, κύριε Μίτσελ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Τον ευχαριστώ που δέχτηκε τις τροπολογίες independent, ανεξάρτητο το λέω αυτό για να κάνουμε ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ του εξαρτώμενου να μην είναι λοιπόν εξαρτώμενα τα στοιχεία αυτά ούτε καν να αμφισβητήσει την ανεξαρτησία. Γι' αυτό ακριβώς θέλω να το διασφαλίσω εν ώψη όλων αυτών που έχουν συμβεί και χαίρομαι ιδιαίτερα που το δεχτήκατε. Όσον αφορά τώρα τα χαμηλά επιτόκια, όταν έρθω, όταν φτάσουν στην Εστονία, πού θα φτάσουν, εδώ και δυόμιση χρόνια, όταν ήρθε εδώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ε, είχα εκπλαγεί με αυτά που μας είπε, αλλά εν τέλει βγήκα αληθινός. Ήμουν εισηγητής για την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του 2007 και είχαμε ζητήσει από την Κεντρική Τράπεζα ότι θα εξετάσουν αυτό το θέμα. Ξέρω ότι με την Κομισιόν το μελέτησαν. Είναι πολύ δύσκολο πώς να αντιμετωπίσει κανείς τα χαμηλά επιτόκια το παραδέχομαι. Συνήθω αυτό γίνεται για να ελεγχθεί ο πληθωρισμό. στο ευρώ, στην ε, ευρωζώνη ε, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη η εφαρμογή των χαμηλών επιτοκίων. Είχε δύσκολε επιπτώσει και ιδίω επειδή οι τράπεζε ε, έβγαζαν τόσα πολλά χρήματα, ήταν τόσο κερδοφόρε, οι άνθρωποι αγόραζαν ακίνητα κλπ. κλπ. Αλλά ήθελα τώρα εν ώψη αυτή τη κατάσταση να δω τι, σε τι συμπεράσματα κατέληξε η Κεντρική Τράπεζα. Σα ευχαριστώ για την ανοιχτή σας προσέγγιση και είναι πολύ, ε, πολύ καλό να βλέπουμε τι γίνεται μέσα σε όλο αυτό το ε, σκηνικό της, του χάους, της ανακατοσούρας που δεν είναι και τόσο χαόδης όσο πολλοί πιστεύουν. Το θέμα είναι να εξασφαλίσουμε την ε, ορθολογική διαχείριση του ευρώ. Ο κύριος Κλίντς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε θα ήθελα όλες οι εκθέσεις τις οποίες είμαι σκιώδης εισηγητής να είναι τόσο σαφείς μακάρι να ήταν έτσι και τόσο ευκολονόητες, ευνόητες όπως σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την έκθεση. Ε, όταν λοιπόν τίθεται το ερώτημα εάν η Εσθονία είναι ε, έτοιμη να ε, ενταχθεί στην Ευρωζώνη εγώ θα ανέτρεπα την ερώτηση και θα ρωτούσα είναι η Ευρωζώνη έτοιμη να δεχτεί την Εστονία η οποία Εστονία είναι έτοιμη, η Ευρωζώνη τι γίνεται θα έπρεπε όμως να χαιρόμαστε, να χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μια χώρα θέλει να μπει στην Ευρωζώνη, διότι όλοι είμαστε βέβαιοι ότι η Ευρωζώνη, παρόλες τις δυσκολίες και τις τα μεγάλα προβλήματα που περνάει τώρα είναι ένα πρόγραμμα, είναι ε, μια, ένα καθεστώς διαρκείας, ε, δεν είναι προσωρινό. Ε, επίσης, από πολιτικούς λόγους υπάρχουν συνάδελφοι, Μάτα, Ανδρεάσεν, που δεν θέλουν δεν συμφωνούν ε, με την είσοδο αυτή της Εστονίας αλλά δεν νομίζω ότι είναι πολιτικά βάσιμα τα επιχειρήματα. Δεν, στο παρελθόν το κάναμε αυτό για ορισμένε χώρες που δεν πληρούσαν τα κριτήρια. Τώρα όμως δεν πρέπει να το επαναλάβω. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνουμε 17 ε, στο άμεσο μέλλον και να, μην, ε, να δεχτούμε την Εστονία και να είμαστε και ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτό το γεγονός. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Η άλλη σκιώδη ηγητής, ο κ. Σκλούτερ, όχι, δεν θέλει να παρέμβει. Άλλος, τους σκιώδη εισηγητές, παρακαλώ, ε, κάποια άλλα παρατήρηση. Τώρα δίνω το λόγο εν κατακλείδη στον εισηγητή μας και θα ψηφίσουμε αύριο για το θέμα 7. Ο εισηγητής, ε, αυτό που ήθελα να κάνω είναι να ευχαριστήσω τους ε, και ότι ηγητές για τη συνεργασία τους υπάρχει μία λεξούλα που θα Α, που διαγράφηκε νομίζω κατά λάθο, αλλά θα την ξαλαβάλω τη λέξη αυτή που κατά λάθο διαγράφηκε και αύριο θα ψηφίσουμε, προσβλέπουμε μεγάλη χαρά στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Προχωρούμε στο επόμενο θέμα. Είναι εδώ ο εισηγητής του θέματος 8 Αποδοχέ διοικητικών στελεχών στιγμών εταιριών και πολιτικέ αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ο κύριος Ελχαντρούη έχει το λόγο. Uh, oh. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, 84 τροπολογίες υπέβαλαν και πρέπει να πω ότι περισσότερες είναι ιδιαίτερα επικοδομητικές και σίγουρα εμπλωτίζουν και βελτιώνουν την έκθεσή μου. Εννοείται ότι υπάρχουν πολιτικές διαφορές, δεν αποτελεί έκπληξη αυτό για κανέναν. Θα προσπαθήσω λοιπόν ως εισηγητής μέσα στις επόμενες ημέρες με τους κοιόδης εισηγητές να καθίσουμε και να βρούμε ποια είναι τα πιο σημαντικά σημεία πάνω στα οποία να πετύχουμε και κάποιους συμβιβασμούς. Πάντως, γενικά μιλώντας, σίγουρα τη σήμερα ημέρα είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταλήξει και να βγει προς τα έξω με ένα σημαντικό μήνυμα όσον αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Βασικό είναι ότι οι υπερβολικές αμοιβέ ε, μπόνους σε στελέχη εισηγμένων εταιριών είναι κάτι που δεν πρέπει να υπάρχει. Αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί παγκοσμίω όλους, την Ευρώπη, τα κράτη-μέλη και άρα χρειάζεται δράση. Μαζί με τη συνάδελφο Μακάρτη, τη δικιά της την έκθεση, ε, πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε κάτι καλό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τις αποδοχές αυτές και τις βασικές αρχές που πρέπει να ισχύουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Το χρονοδιάγραμμα είναι καλό, γιατί να, μέχρι αύριο περιμένουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει έκθεση για την εφαρμογή των ε, συστάσεων που έγιναν το 2009 για να πει τι έχει γίνει τελικά στα κράτη-μέλη. Από ό,τι έχουμε ακούσει, χρειάζεται ακόμα δουλειά. Ότι η κατάσταση χρειάζεται μεγαλύτερη δουλειά. Δεν έχουμε δηλαδή τα αποτελέσματα που περιμέναμε εντελώς. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύριο θα μας δώσει και την ε, πράσινη βίβλο της για το δημοσιονομικό τομέα όπου θα ζητάει πιο αυστηρές διαδικασίες εσωτερικά και από ό,τι έχω καταλάβει εγώ μπορούμε να περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του 2011 να έχει ετοιμάσει ένα πλαίσιο για τον δημοσιονομικό τομέα και για τις εισαγμένες εταιρείε στο χρηματιστήριο. Τώρα όσον αφορά τις τροπολογίες. Δεν θα μπω βέβαια σε λεπτομέρειες για όλες αυτές τις τροπολογίες, αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα με τα οποία συμφωνώ. Για παράδειγμα, της συναδέλφου Βότμαν Κόλ για το Ταμείο Κρίσης. Νομίζω ότι διατυπώνεται πολύ καλά. Υπάρχουν επίσης ορισμένοι οι οποίοι θέλουν κάποια αναλογικότητα και εδώ συμφωνώ. Η τροπολογία 67 που μιλάει για τις αμοιβέ όχι μόνο για τους μισθούς αλλά και για τις συντάξεις. Το σύνολο ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Όντως πρέπει να διευκρινιστεί αυτό. Επιπλέον πέρα από διάφορους συμβασμούς που σας είπα που θα τους καταφέρουμε στο τέλος, παραμένουν και κάποιες διαφορές μεταξύ μας. Νομίζω ότι είναι σημαντικό η διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων από μια εταιρεία ε, πρέπει να περνά από έγκριση, από κάποια εποπτεία. Δηλαδή η ιδέα πρέπει να είναι ότι η εταιρεία μπορεί να οργανωθεί, πρέπει να έχει τη δομή, τις διαδικασίες που χρειάζεται για να μπορεί να τα βγάλει πέρα με τους κινδύνους. Και σε αυτό πρέπει βέβαια να μπορεί να την ελέγχει κάποιος απ' έξω. Οπότε, χαίρομαι εδώ για την στήριξη της κυρίας Μπόρς. Επίσης, είμαι πεπισμένος ότι ο ρόλος του επόπτη πρέπει να βγαίνει ενισχυμένος από την έκθεση η ισορροπία ανάμεσα στον κίνδυνο και τις αμοιβέ και εδώ πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία. Και τέλος εγώ λέω ότι πέρα από τα αναφέρει η έκθεση Μακάρδη για τις αγμένες εταιρείε ότι και για αυτές πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία και κάποιες συμφωνίες με διαφάνεια όσον αφορά τους μισθούς, τις αμοιβέ. Κάποια άλλα πράγματα τα οποία μπορούμε να διαπραγματευτούμε είναι την αναλογία ανάμεσα στη, στο μεταβλητό σκέλος και το σταθερό σκέλος των αμοιβών. Και από αυτού θα κάνω μια πρόταση. Επίσης υπάρχουν συνάδελφοι που πιστεύουν ότι δεν πρέπει να λέμε αρκετά περισσότερα πράγματα για τις αμοιβέ, άλλοι που λένε ότι πρέπει να πούμε ακόμα περισσότερα, για περιορισμό των αμοιβών δηλαδή. Αλλά βλέπετε με την κρίση που έχουμε τον τελευταίο χρόνο τα πράγματα πρέπει να εξελίσσονται έτσι που να είναι υπεύθυνα. Γι' αυτό αξίζει τον κόπο να τα συζητήσουμε για να μην πάρουν ανακατήφορο χωρί τέλο. Τώρα από εδώ και πέρα θέλω να ακούσω τις αντιδράσεις των συναδέλφων. πρέπει να δούμε μαζί τι βελτιώσεις μπορούμε να επιφέρουμε στην έκθεση αυτή τελικά και μετά θα ψηφίσουμε, έτσι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Νίτσας. Ευχαριστώ. Πρέπει να τονίσουμε ένα θετικό στοιχείο αυτής της έκθεσης Και αυτό είναι η διασύνδεση μεταξύ αμοιβών και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων. Πρέπει η Επιτροπή η οποία κρίνει τις αποδοχές να είναι ανεξάρτητη και αντικειμενική. Σε αυτό υπάρχει πιστεύω ε, συνένεση απόψεων και εφόσον συναντηθούμε με τον εισηγητή για να το συζητήσουμε ε, θα ρωτούσα εάν πιστεύει ότι οι αποδοχές είναι το βασικό αίτιο της κρίσης. Εδώ έχω ορισμένε αμφιβολίες. Είναι ένας παράγοντας που συνέβαλε στην ε, τεράστια κρίση, αλλά όχι ο μόνος όχι μοναδικός. Εάν δούμε τώρα τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί ε, για την ε, φορολόγηση, την επιβολή ε, φόρου, η φορολόγηση υπερβολικών αποδοχών δεν είναι δεν εφαρμόζεται στην Ευρώπη, ούτε πιστεύω υπάρχει γενική αποδοχή μιας τέτοιας προσέγγισης. Θα ήμουν ευτυχής να ακούσω την άποψη του εισηγητή για αυτή την επιβολή φόρου, για αυτή την ιδέα επιβολής φόρου, αλλά δεν βλέπω ποια δικλίδα ασφαλείας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αποφύγουμε μια μελλοντική παρόμοια κρίση. Αυτή η ιδέα λοιπόν της επιβολής ενός φόρου σε υπερβολικές περιπτώσεις δεν νομίζω ότι είναι εφικτή, δεν, δεν είναι ρεαλιστική. ο βασικός στόχος, η βασική κατεύθυνση που ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σωστή. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε μία μονάδα επαφής, μία μονάδα ανταλλαγής πληροφοριών αντί μίας ε, ε, ανεξάρτητης επιτροπής ε, ελέγχου και παρακολούθησης των αποδοχών. Πρέπει να δούμε καταρχάς τι έχει επιτύχει το παρόν ρυθμιστικό πλαίσιο και πώς έχει επηρεάσει τις αποδοχές. Έχει το ρυθμιστικό πλαίσιο επηρεάσει θετικά την εξέλιξη των αποδοχών ή είχε αρνητικά, αρνητικές επιπτώσεις. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Γενικά και εγώ με μεγάλο ενδιαφέρον θέλω να συζητήσω το θέμα αυτό με τον εισηγητή. Όπως ο κύριος Νίτρας είπε μόλις τώρα, συμφωνώ με την προσέγγιση του πολλά ιδέες έχουν ακουστεί για το πώς μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση, τι μέτρα μπορούμε να εφαρμόσουμε, ε, ίσως να εφαρμόσουμε νέα μέτρα σε αυτό το πεδίο και οι, επίσης ορισμένες επικρίσεις για μέτρα που εφαρμόστηκαν και ήταν, δεν ήταν ικανοποιητικά. Ας μην ξεχνάμε και την αναλογικότητα. Υπάρχουν διαφορετικές επιχειρήσεις. Ε, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τα ίδια στους πάντες. Δεν, δεν, δεν είναι λογικό ε, αυτό. Επίσης, ας, μη, ας θυμόμαστε ότι η Ευρώπη δεν είναι μια φούσκα. Ε, οι παν, παγκόσμιες αποφάσεις που έχουν ληφθεί ας πούμε από τους G20 είναι πολύ σημαντικές ως βάση να έχουμε υπόψη μας το πλαίσιο αναφοράς των αποφάσεων των G20 για να δούμε και να κρίνουμε τι γίνεται παγκοσμίω. Ορισμένες από τις τροπολογίες θέλουν να ενισχύσουν τους μετόχους πρέπει να έχουμε μια πολύ προσεκτική προσέγγιση και να είμαστε πολύ σοβαροί ε, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ μερισμάτων και αποδοχών. Δεν νομίζω ότι οι συνδικαλιστικοί φορείς πρέπει να ανακατευθούν ή έχουν κάτι να κάνουν ε, σε αυτό το πεδίο. Γενικά δεν έχω πιστεί ότι εμείς ως πολιτικοί μπορούμε να παρέμβουμε και να θέσουμε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία και ποσοστά για τις αμοιβέ ε, και να τα υποβάλουμε αυτά αυτά ως τροπολογίες. Δεν μπορούμε να είμαστε υπερβολικά συγκεκριμένοι. Επίσης, ε, Μην, μην ξεχνάμε ότι πολλές από τις αποδοχές και τα bonuses κρίνονται από τις εταιρείες τις ίδιες που αξιολογούν τις αποδόσεις των στελεχών τους. Γι' αυτό πρέπει να δούμε εάν μπορούμε να εφαρμόσουμε μια γενική προσέγγιση η οποία να είναι αναλογική ε, σε όλες τις εταιρείες Εγώ πιστεύω πριν υιοθετήσουμε νέα μέτρα ή πριν λάβουμε νέε αποφάσει πρέπει να αξιολογήσουμε τα μέτρα τα οποία έχουν εφαρμοστεί, έχουν ληφθεί μέχρι τώρα και να προσέξουμε να κάνουμε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση πριν εγκρίνουμε νέου ρυθμιστικού φορεί και ε, ζητήσουμε την επιβολή νέων μέτρων νέων φορέων δηλαδή εποπτείας και παρακολούθησης. Ας κάνουμε μια σωστή αξιολόγηση της εξέλιξης των αποδοχών και των επιπτώσεων των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα. Και προσβλέπω και εγώ με μεγάλη χαρά στη συζήτηση αυτή που θα γίνει με τον εισηγητή. Η κυρία Φόρντ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον εισηγητή για την εργασία του πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλές συμφωνίες για την πολιτική προσέγγιση των αποδοχών διεθνώ και χρειάζονται, χρειάζεται ένα στεναρό πλαίσιο ρυθμιστικό. Πρέπει όμως να είμαστε σαφείς σχετικά με την ε, επέκταση με τη διεύρυνση των μέτρων αυτών εκτός του ε, χρηματοοικονομικού τομέα όπου δεν υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες. Ε, εάν θέλουμε η προσέγγιση μας να υπερβεί το χρηματοοικονομικό τομέα, πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα ζημιωθούν όσον αφορά τη διεθνή τους ανταγωνιστικότητα. Συμφωνώ με αυτά που είπε μόλις ο Κάρλ. Θα πρέπει αναλογικά να δούμε τι μπορούμε να εφαρμόσουμε σε ποιον για να μην θυγούν αρνητικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι άλλες μικρότερες επιχειρήσεις οι οποίες ε, δεν έχουν τη δυνατότητα να να εισάγουν μία ανεξάρτητη ε, επιτροπή αξιολόγησης των αποδοχών. Λοιπόν, πρέπει να δούμε και την ποσοτική αξιολόγη, ε, αναλογικότητα των επιχειρήσεων όσον αφορά τα μεγέθη τους και το θέμα των μετόχων, της ευθύνης των μετόχων. Ε, πρέπει και αυτή η ευθύνη των μετόχων να μελετηθεί όσον αφορά δε τους εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελέγχους και αυτό να το εξετάσουμε όπως επίσης και τους, τα διευθυντικά στελέχη χωρίς εκτελεστική εξουσία. Και αυτόν, αυτόν τον ρόλο ε, πρέπει να δούμε. Ίσως ε, μπορούμε να εφαρμόσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο για, τους για τα μη εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη της χώρας μου και σε άλλες ε, περιπτώσεις. Ε, ας μελετήσουμε και την έκθεση του ΩΣΑ για τις αποδοχές. Αναφέρει τη σύνδεση μεταξύ της ανάληψης κινδύνου και των αποδοχών. Εδώ υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Όταν ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αξιολογεί κινδύνους, τους οποίες ε, θέλει να διατηρήσει για το δικό του ισολογισμό, τότε οι φορείς, ήδη το άτομο ή οι, οι αρχές οι οποίες εγγυώνται το ρίσκο αυτό, ε, προτιμούν το ρίσκο αυτό να κατανεμηθεί σε διάφορους άλλους. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Ε, πολλές φορές ένα το, το, το, ο κίνδυνος το οποίο αναλαμβάνει ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ε, μπορεί να ε, είναι διαφορετικό, να κατανέμεται διαφορετικά και να μην είναι κατάλληλο για ένα συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ενώ να είναι κατάλληλο για άλλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς ήθελα να σημειώσετε ότι εδώ έχουμε μια πρόταση η οποία προσεγγίζει ιδιαίτερα το αμερικανο-βρετανικό σύστημα, το επιχειρησιακό σύστημα το οποίο διαρρείται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη. Στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο Έχουμε μία ε, διοικητική, ε, ε, έχουμε δύο βαθμίδες στη διοίκηση των επιχειρήσεων. Και πιστεύω ότι αυτή η δυνατότητα των δύο βαθμίδων πρέπει να διατηρηθεί. Τώρα, εάν ασχοληθούμε με τις αποδοχές των directors, των διευθυντών, των διευθυντικών στελεχών, τότε δεν συμπεριλαμβάνουμε όλους αυτούς οι οποίοι τουλάχιστον στα μάτια της δημοσιότητας λαμβάνουν υπερβολικές αμοιβέ. Παραδείγματο χάρη στην Deutsche Bank ο Γιώζεφ Άκερμαν, ο, ο διευθυντής, ο γενικός διευθυντής παίρνει 11 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο αλλά ε, είναι στον κατάλογο των καλύτερων ε, πληρωμένων στελεχών της Deutsche Bank στο νούμερο 70 ή 80. Δηλαδή ο άνθρωπος παρόλο το μισθό που παίρνει είναι 70 στη σειρά μεγέθους αποδοχών. Ε, Ενώ υπάρχουν ε, traders και brokers οι οποίοι κερδίζουν πολλαπλάσια από το Γιώζεφ Άκερμαν. Άρα λοιπόν το πρόβλημα αυτό δεν λύνεται έτσι και ο Καρλ ήδη το είπε. Ως μέλος μιας φιλελεύθερης ομάδας Ήδη μου πέφτει δύσκολο να δεχθώ ότι η πολιτική θα παρέμβει στις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων. Εμείς ε, έχουμε ρυθμιστική αρχή επιθεώρησης, έχουμε ε, μια γενική συνέλευση μετόχων ε, μέσα στο νομοθετικό μας πλαίσιο. Έχουμε μια εταιρική, ένα εταιρικό σώμα διακυβέρνησης. Πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι φορείς εντός των επιχειρήσεων που ορίζονται από την νομοθεσία επαρκούν, φτάνουν εντάξει δεν λέω ότι μπορούμε ε, κάτι να κάνουμε αλλά να μην γελιόμαστε ας απο... ό,τι και να αποφασίσουμε αν κάποιος θέλει να παρακάμψει τις αποφάσεις μας ή να βρει παρασυράκια θα τα βρει ε, το είδαμε αυτό και πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, σκέφτηκαν εφαρμόσουν έναν φόρο για τα bonuses, για τα πριν που παίρνουν, τα μεγάλα πριν των τραπεζών, άρχισαν αμέσω να βρίσκουν ε, ε, μέτρα διαφυγής, ε, πώς να ξεφύγουν δηλαδή τα στελέχη από το φόρο αυτό, τον ενδεχόμενο. Δεν θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε το λάθος να ορίσουμε ορισμένους ποσοστά να πούμε ας πούμε ότι 50% του μπόνους θα φορολογηθεί θα το πάρει ο φόρος Αλλά πρέπει ταυτόχρονα να μην ξεχνάμε ότι αυτή η τεράστια μισθή είναι πέραν κάθε μέσου όρου. Πώς θα εξηγήσουμε σε έναν μικρό μεσαίο άνθρωπο ότι ότι ο υπεκεφαλής γιατρός ενός νοσοκομείου κερδίζει 80.000 ευρώ με την εμπειρία που έχει, ενώ ένας χρηματιστής κερδίζει 80 εκατομμύρια ευρώ. Πώς θα τα εξηγήσουμε αυτά στον απλό άνθρωπο. Ε, ό,τι όμως και να αποφασίσουμε πιστεύω ότι πρακτικά δεν θα αλλάξουν πολλά. Η πραγματικότητα υπερβαίνει τις ρυθμίσεις. Έχω συμφωνώ με το περιεχόμενο, με την ουσία της έκθεσης και την μακροπρόθεσμη και την μεσοπρόθεσμη προσέγγιση. Εάν αποφασίσουμε και θέλουμε να παρέμβουμε, τότε θέλουμε να συμπεριλάβουμε, πρέπει να συμπεριλάβουμε όλους τους εργαζόμενους, όλα τα στελέχη μιας επιχείρησης που έχουν γιγαντιές απολαβές. Και εγώ δεν καταλαβαίνω πραγματικά γιατί ένα τέλεχο τη Deutsche Bank κερδίζει 12 εκατομμύρια ευρώ το, χρόνο. εμφανιζόμενο, εμφανιζόμενος σποραδικά στην, ε, ε, στη δουλειά του. Ε, δεν λέω ότι πολλά άσχημα συμβαίνουν, αλλά ας προσέξουμε την ουσία. Εγώ έχω να κάνω κάποια σχόλια. Το μικρόφωνο σας είναι ακόμα αναμένα. Μάλιστα, ευχαριστώ. Το σχόλιο που εγώ θέλω να κάνω είναι ότι πιστεύω πως είναι σωστό και αναφέρθηκε ήδη ότι στόχο θα πρέπει, στόχος θα πρέπει να είναι αναλογικότητα. Και όταν θα συντάξουμε τις ε, συμβαστικές τροπολογίες, αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Οι δικές μου τροπολογίες βασικά είχαν στόχο να προσπαθήσουμε να έχουμε έναν κάποιο βαθμό συμφωνίες ανάμεσα στην προσέγγιση που ακολουθούμε εδώ και την προσέγγιση που ακολουθούμε στην οδηγία για τις απαιτήσει ε, κεφαλαίου. Ίσως θα πρέπει κάπως να τα ξαναδούμε για να δούμε σε ποιο επίπεδο μιλάμε. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να ασχοληθούμε με την μεγάλη δυσαναλογία των τεράστιων πριμ που δίνονται, που μπορεί να στρεβλώσουν τα πράγματα αν ε, αυτό αφορά τη ε, πάνω στρώματα της ε, καθετερίας και στην οδηγία περί απαιτήσεων κεφαλαίου θα πρέπει και αυτό να το συζητήσουμε αντίστοιχα με τα ποσά που κερδίζουν και θα πρέπει να θα το δούμε αυτό σε λίγο Άκουσα τόσο, είπε ο Βόλφ για το ότι ό,τι και αν κάνουμε θα, ο κόσμος θα προσπαθεί να τα παρακάμψει, αλλά δεν νομίζω πως αυτό είναι λόγος να τα καταλήψουμε την προσπάθεια. Και σίγουρα, αν είναι γνωστό από τους ε, μετόχους ποια είναι η πρόθεση της νομοθεσίας, αυτό δίνει περισσότερο βάση στους ε, μετόχους αν πάνε σε μια συνεδρία των μετόχων και πούν ότι μπορεί εντάξει να μην ε, τηρήσεις απόλυτα την νομοθεσία αλλά ε, να προσπαθήσεις να την παρακάμψεις. Αυτός δεν είναι λόγος για να μην προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι και ίσως και τα ίδια τα κράτη-μέλη θα είναι αρκετά έξυπνα στον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσουν όλα αυτά. Τέλος, για τα κονδύλια διάσωσης έχουμε μία πρόταση από την Κομισιόν για ένα τέτοιο ταμείο που βοηθά στην, στο κλείσιμο μιας εταιρείας και δίνει ε, κάποιο κεφάλαιο λειτουργικό αν έχει να κάνει κανείς με μια διασυνοριακή πτώχευση ε, μπορούμε αυτά να έχει κάποιες ενδιαφέρουσες ιδέες για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την διασυνοριακή μεταφορά, έμβασμα μάλλον, αν υπάρχει μια διασυνοριακή, ένα διασυνοριακό θεσμό, ανήκει ας πούμε σε ένα κράτος μέλος, αλλά λέει το εποπτικό όργανο ότι δεν φεύγουν χρήματα από τη χώρα μου που επειδή πρόκειται μόνο για ακίνητες περιουσίες και να μπορούν να το παρακάμψουν Και ίσω εκεί θα πρέπει να μπορούν να το εξετάσουν περισσότερο, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να υιοθετηθεί ως γενική λύση που θα προσπαθούμε να την εφαρμόζουμε σε κάθε περίπτωση. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να είμαστε βέβαιοι πω θα έχουμε του σωστού κανόνε για να αντιμετωπίσουμε την διασυνοριακή αφεργιότητα. Και δεν νομίζω πως αυτή είναι η έκθεση εντός της οποίας θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Αυτά. Και Και έχω και τον κύριο Κρούτρ και μετά τον εισηγητή. Εντάξει, ο κύριο Κρούτ πρώτα. Ήθελα κι εγώ ε, να ευχαριστήσω τον εισηγητή καταρχάς. Μια πάρα πολύ χρήσιμη έκθεση Συμφωνώ όμως μετά από αυτά που είπε ο κύριος Κλίντς δεν έχει άδικο σχετικά με το, τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει στις αποδοχές μεταξύ αυτών που πραγματικά παράγουν, κάνουν κάτι χειροπιαστό στη δουλειά τους, που παίρνουν πολύ, λιγότερο, πολύ λιγότερα χρήματα από τη δουλειά τους και αυτούς οι οποίοι είναι στα υψηλά ε, ε, στους ψηλούς ορόφους και μαζεύουν ε, πάρα πάρα πολλά. Αυτή η ψαλίδα λοιπόν είναι τεράστια και πιστεύω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Τουλάχιστον είναι η αρχή αυτή της προσπάθειας. Ορισμένες τροπολογίες, ιδιαίτερα του Πασκάλ, ε, υποστηρίζω, τις θεωρώ λογικές, αλλιώς ε, πιστεύω ότι η έκθεση είναι καλύτερα στην αρχική της μορφή και δεν βελτιώνεται με τις τροπολογίες. Προτιμώ την έκθεση στην αρχική της μορφή. Ευχαριστώ. Okay, thank you. Um... Ωραία, σας ευχαριστώ. Βλέπω που έρχεται ο κύριος Κάντερ. Τώρα συζητάμε τι τις ε, αποδοχές των ε, διευθυντών ε, εγγεγραμμένων εταιριών, η Αρλίν. Εγώ δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα υπόθηκαν. Φυσικά και υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στι δύο οδηγίε και εκτιμώ τη δουλειά του εισηγητή. Είναι σημαντικό, όπω είπαν και διάφοροι άλλοι, η Επιτροπή να ηγηθεί σε αυτά τα θέματα, γιατί νομίζω πω το κοινό είναι στραμμένο προ εμά εδώ ω νομοθέτε, όχι για να λάβουμε απόφαση για το πόσα θα πρέπει να πληρώνει το καθένα, αλλά για να θεσπίσουμε ένα πλαίσιο, ένα γενικό πλαίσιο, γιατί μιλάμε για ένα κλάδο που έχει ξεφύγει Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε, ε, να, να αμφισβητήσουμε αν ένας πούμε, θα πρέπει να παίρνει 4 εκατομμύρια το μήνα ή αν ε, ένα φωτομοντέλο θα πρέπει να παίρνει τα, ε, κάποια, κάτι αντίστοιχο και ούτω καθεξής. Μα δεν είναι δικά μας χρήματα. Εδώ μιλάμε για κινδύνους, για ανάληψη κινδύνων και μιλάμε για κόσμο ο οποίος καταθέτει στην τράπεζα και κινδυνεύει να χάσει τα χρήματά του λόγω αυτών των μισθών. Εμεί δεν καθορίζουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με αμοιβέ αποδοχές ε, στι ε, εταιρείε, ε, εκτός όταν αυτό φτάνει σε υπερβολικά ύψη. Δεν ήταν το αίτιο της κρίσης, αλλά η υπερβολική ανάληψη κινδύνου ήταν τμήμα της κρίσης. Δηλαδή ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν έτοιμοι να αναλάβουν τεράστιου κινδύνους ώστε να έχουν μεγάλα κέρδη και αυτό συνέβη. Υπάρχει άμεση σύνδεση λοιπόν ανάμεσα στις πολιτικές αμοιβή ε, και την ε, τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Και συμφωνώ με τους συναδέλφους που λένε ότι φυσικά θα πρέπει να κινηθούμε σε διεθνές επίπεδο βήμα προς βήμα σε αυτό το τομέα, αλλά αν δούμε αυτές τις αρχές σαφώς ε, είναι, φαίνεται ότι είναι απαραίτητο να έχουμε μια, πιο αναλογική ε, και πιο ισορροπημένη προσέγγιση στον ε, χρηματοπιστωτικό τομέα. Γιατί διαφορετικά γιατί φτιάχτηκε αυτό το γραφείο ε, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας θα μπορούσε ας πούμε ένας εργαζόμενος να κερδίζει το δικό του μισθό από το 90%, το 90% μάλλον του μισθού του να είναι ένα πριμ. Ε, είναι και αυτή μια ιδέα και ήμουν ευτυχής που είχαμε την ευκαιρία ε, με την έκθεση CRD ε, τρία είχαμε μια συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής της Βασιλείας και είπε συγκεκριμένα πως οι τράπεζες θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις κεφαλαίων τους αν δεν πλήρωναν τόσο τεράστια ποσά ε, ως πριν. Η κουλτούρα λοιπόν αυτού εδώ του κλάδου είναι και έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε τα προσωπικά κέρδη να είναι, να είναι πιο σημαντικά από την υγεία του ίδιου του θεσμού. Μα είπε επίση ότι 40% των πλονασμάτων ε, τη εταιρεία ε, το έβγαζαν από το κεφάλαιο και αυτό έχει να κάνει με την υγεία των χρηματοπιστωτικών αυτών ιδρυμάτων. Έχουμε λοιπόν νομοθετική υποχρέωση και καθήκον να θεσπίσουμε κάποιου κανόνε σε αυτό το τομέα. Χωρί βέβαια να τα λέμε όλα με τον ή και με το σίγμα, αλλά και να δίνουμε και κάποιο βαθμό ευελιξία. Να μην υπερβάλλουμε δηλαδή όσον αφορά την υποβάθμιση, τον αρνητικό αντίκτυπο σε μικρότερα θεσμικά όργανα. Και βέβαια να κάνω και το ίδιο σχόλιο όπως και η Επίτροπος για το σχόλιο, η Πρόεδρος στο σχόλιο του κ. Κλίντς, ότι όντως αν εμείς ρυθμίζουμε και αν νομοθετούμε, ο κόσμος πάντα βρίσκει τρόπο για να παρακάψει να βρει παραθυράκι. Αλλά δυστυχώς δεν είναι αυτό φοβερό ε, για έναν κλάδο που δεν έχει αλλάξει. Ε, δηλαδή προσπαθεί να παρακάμψει διαρκώ την νομοθεσία ώστε να συνεχίσει αυτή την πρακτική των αμοιβών. Ενώ σαφώ δεν είναι αποδεκτό κάτι τέτοιο για τον κόσμο. Και για όσους πιστεύουν ότι χρειάζεται να γίνουν αλλαγές σε αυτό το τομέα, το χρηματοπιστωτικό. Εγώ νομίζω ότι πρέπει κάτι να κάνουμε να, δεν μπορούμε να λέμε ότι επειδή οι άλλοι θα βρουν παραθυράκια ότι δεν πρέπει εμείς να κάνουμε τίποτα και ο κύριος Κλίντ συγκεκριμένα ανέφερε το Ηνωμένο Βασίλειο. Και να σας πω ότι το Υπουργείο Οικονομικών κατέστησε σαφές στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ότι δεν πρόκειται να τους αφήσουν να βρουν παραθυράκια και ότι θα προσλάβει δικούς του δικηγόρους ώστε να δει τι είδους παραθυράκια θα μπορούσαν να προβλεφθούν. Γι' αυτούς τους λόγους ακριβώς θα πρέπει να στηρίξουμε τις συστάσεις στην έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω το λόγο, οπότε δίνω το λόγο στον εισηγητή πάλι για να απαντήσει στα διάφορα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τους συναδέλφους. Πρέπει να δούμε πώς πάνε τα πράγματα σήμερα θα μπορούσε να πει κανείς. Να περιμένουμε λίγο, να μην υπερβάλλουμε, αλλά στην πραγματικότητα εγώ πιστεύω ότι αυτά που θα δημοσιευθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύριο για τις συστάσεις του Ιουνίου του 2009, κατά πώς έχουν τεθεί σε εφαρμογή δηλαδή και πώς, εκεί θα λέει ότι τα κράτη-μέλη τελικά δεν έχουν εφαρμόσει τις συστάσεις αυτές. Και ότι εξακολουθεί να ισχύει το σύστημα των υψηλών αποδοχών στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θέλω να επιμείνουμε στις συστάσεις αυτές. Επίσης, αυτό το θέμα πρέπει να το δούμε κάπως γενικά και να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που θα περιορίσουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό για να περιορίσουμε τις δυσκολίες. Πάντως συμφωνώ με εκείνους που λένε ότι δεν πρέπει να περιορίσουμε μόνο τις αποδοχές των πολύ ψηλά εσταμένων, γιατί υπάρχουν και άλλοι που είναι πιο κάτω, που και αυτοί κερδίζουν πάρα πολλά, που και αυτοί διαχειρίζονται κινδύνους κατά κάποιο τρόπο. Ναι, είναι αλήθεια. Και με ορισμένες τροπολογίες αυτό γίνεται. Πάντως, όπως είπα και στην αρχή, θα καθίσουμε με τους σκιώδεις εισηγητές να δούμε πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε και σίγουρα θα παίξει ρόλο και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιμένουμε αύριο. Οπότε εκεί θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε εμείς ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή και γενικότερα ως Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Οπότε θα ψηφίσουμε στις 22 Ιουνίου εδώ στην Επιτροπή μας και τον Ιούλιο θα πάει η έκθεση αυτή για ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Συνεχίζουμε τώρα και περνάμε στο τελευταίο θέμα για σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Εκτός αν προκύψει κάτι άλλο, δεν ξέρω. Και αυτό είναι να δούμε τις αγορές παραγόγων, μελλοντικές δράσεις πολιτικής. Έκθεση του Βέρνερ Λάγκεν. Οπότε θα δώσω το λόγο στον εισηγητή πρώτα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχουμε πολλές φορές συζητήσει την έκθεση και τις τροπολογίες. Εγώ προσπάθησα να βρούμε μία όσο το δυνατόν ε, ενιαία ομοιόμορφη ρύθμιση στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν οι περισσότεροι συνάδελφοι. Οι συμβιβαστικέ ε, τροπολογίες τις συζητήσαμε τις τελευταίες δέκα μέρες ε, ενδελεχώς και σε διμερές επίπεδο και σε επίπεδο πολιτικών ομάδων. Πιστεύω λοιπόν ότι με το συνδυασμό αυτό επιτύχαμε καθαρά, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε τη γραμμή που θέλουμε να ακολουθήσουμε όσον αφορά την ομοθεσία και από την άλλη τις διαφορές ε, των απόψεων ε, που υπάρχουν για τα παράγωγα. Οπωσδήποτε τα παράγωγα είχαν μία έντονη ε, επίπτωση στις χρηματοοικονομικές αγορές, όμως τελικά ε, έχουν μία πολύ αμφιλεγόμενη θέση όσον αφορά την διασπορά του κινδύνου. Ε, έχουμε λοιπόν τα εκτιμώντας, καταρχάς τα πρώτα 8 εκτιμώντας και εν συνεχεία μέχρι την τροπολογία 21 Ε, έχω ενσωματώσει πολλές προτάσεις, πο, πολλές ιδέες ε, σε, αυτά, σε αυτά ε, τις πρώτες τροπολογίες και σε αυτά που αφορούν τα εκτιμώντας. Οι σοσιαλδημοκράτες, η ΠΕΠΕ, το ΕΛΚ, οι πράσινοι και οι φιλελεύθεροι έχουν υποβάλει τροπολογίες. Εγώ όπως σας είπα προσπάθησα να επιτύχω, να, να εφαρμόσω μια ανοιχτή προσέγγιση έτσι ώστε να μπορέσει να περάσει η έκθεση αυτή με όσο το δυνατό μεγαλύτερη πλειοψηφία. Γι' αυτό δεν ε, ε, ε, εστίασε την προσοχή μου σε συγκεκριμένε λέξεις ή σε αριθμού τροπολογιών. Εγώ ήθελα να περάσει όσο το δυνατόν μια ομοιόμορφη γραμμή διαμέσου του Κοινοβουλίου που να εκφράσει στεναρά τι απόψεις μα όσον αφορά τα παράγωγα. Τα εκρεμή ζητήματα, τα επίμαχα ζητήματα είναι, αν αρχίσουμε από τα εκτιμώντας, συμφωνώ ότι τα παράγωγα παίζουν ένα χρήσιμο ρόλο κλπ. κλπ για τις οικονομικές αγορές, όμως ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές σύμφωνα με τη φύση του προϊόντος ε, και ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές όσον αφορά τη ρύθμιση και τη διαφάνεια και ότι έχουν παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την, ε, στην οικονομική αυτή κρίση. Τι... Λοιπόν, α, είχα κάποια... κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Λοιπόν, ε, τροπολογία 1 ε, αφορά το εκτιμώντας 7. Όλοι έχουν συμφωνήσει σε αυτό. Η τροπολογία 2 αφορά την, το εκτιμώντας 7α. Ε, Ε, ε, εστιάζεται στις αδυναμίες της αγοράς παραγόγων και εδώ έχουν συμφωνήσει όλοι. Ε, τροπολογία συμβιβαστική 3 είναι 26, είναι τροπολογία 26 της κυρίας Ποδηματάς της κυρίας Ποδηματά η οποία την έχω διαιρέσει σε τρία τμήματα και θα ψηφιστεί λοιπόν ξεχωριστή, ψηφοφορία. Στο δεύτερο τμήμα προτείνω αρνητική, δηλαδή καταψήφιση. Στο πρώτο τμήμα υπερψήφιση, στο δεύτερο καταψήφιση. το δεύτερο μέρος αναφέρεται στις αρνητικές επιπτώσεις των παραγόγων και πώς έχουν ε, ε, διακυβεύσει όλη την υποδομή της Ευρωζώνης. Εδώ λοιπόν δεν συμφωνώ ε, δεδομένου ότι σε ορισμένες φορές τα παράγωγα είχαν αρνητική ή θετική επίπτωση. Στην περίπτωση της Ελλάδος που, όπου έχουμε τα στοιχεία 310 δισεκατομμύρια δάνεια, είχαμε όμως μία ασφάλεια αθέτησης αποπληρωμής 6 εκατομμύρια ευρώ, ε, δισεκατομμυρίων ευρώ, που ε, αν το πολλαπλασιάσουμε επί 12,5 έχουμε 75 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου ένα τέταρτο του συνολικού ελληνικού δανείου ε, καλύπτεται από ασφάλεια σε περίπτωση αθέτησης αποπληρωμής του χρέους, ε, σε περίπτωση κινδύνου αθέτησης υποχρέωσεων. Γι' αυτό θα ήθελα το μεσαίο τμήμα να το διαγράψουμε από την τροπολογία της κυρίας Ποδηματά υπαρθμών 26 και να κρατήσουμε το πρώτο και το τρίτο μέρος. Εν συνεχεία έχουμε τη συμβαστική τροπολογία 4 που υποστηρίζεται από τις πέντε ομάδες. Ε, που αναφέρεται στο εκτιμώντας α και αναφέρεται στην επιθυμία της Κομισιόν για αυστηρότερη ρύθμιση, ε, ρυθμιστικό πλαίσιο. Συμφωνώ σε αυτό. Συμβιβαστική τροπολογία 4 για ξεχωριστή ψηφοφορία. Αυτό το ζητάει, το ζητούν οι σοσιαλδημοκράτες, πράσινοι, Άλτε, έλκ ε, και συντηρητικοί. Ε, πρώτο και δεύτερο τμήμα. Το δεύτερο τμήμα λέει ότι ορισμένα παράγωγα χρησιμοποιήθηκαν για κερδοσκοπικούς σκοπούς και θα πρέπει να υπόκεινται σε ε, ρυθμιστικό πλαίσιο. Ε, η συμβιβαστική τροπολογία 5 είναι αυτή ε, που αναφέρεται στο εκτιμώντας G. για το δεύτερο τμήμα έχουμε μία πρόταση των σοσιαλδημοκρατών που ζητούν ξεχωριστή ψηφοφορία. Εγώ πιστεύω ότι η επιχειρηματολογία είναι σωστή αυτή τη τροπολογία του δεύτερου τμήματος, όμως δεν έχουμε επιτύχει συμφωνία, οπότε θα γίνει ξεχωριστή ψηφοφορία. Προχωρούμε στο, ε, τελευταίο ε, εκτιμώντας H, είναι η συμβαστική τροπολογία 6, ε, κατόπιν αιτήματος των σοσιαλδημοκρατών που λέει ότι υπάρχει συστημικός κίνδυνος όσον αφορά τον όγκο των συναλλαγών τον οποίο αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει ο τελικός χρήστης. Οι συμπληρώσεις που συζητήθηκαν εχθές και υποβλήθηκαν, ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί στις 10 στη Γενική Γραμματεία δεν έχω συμπεριληφθεί στη συμβαστική τροπολογία αλλά θα έγιναν δεκτές ως προφορικές τροπολογίες. Ξέρουμε ότι υπάρχει εδώ ποιοτική διάκριση. Εγώ θα ήθελα να είχαν συμπεριληφθεί στις, προφορικές τροπολογίες, στις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες, διότι όταν υποβληθούν προφορικά δεν μπορούν να, να, ψηφιστούν και παρακαλώ τη γραμματεία να συμπεριληφθεί ε, αυτό το σημείο στη συμβιβαστική τροπολογία παρόλο που ε, υποβλήθηκε σήμερα το πρωί στις 10. Αύριο θα το ψηφίσουμε. Έχουμε ακόμα περιθώριο, μπορούμε να αλλάξουμε στις συμβιβαστικέ τροπολογίες. Και επίσης ε, σας παρακαλώ να αναγνωρίσετε την ποιοτική διάκριση που, που υπάρχει και να μην επιτρέψουμε ε, ακριβώς τον κίνδυνο της κερδοσκοπίας. Συμβιβαστική τροπολογία 7 εδώ υπάρχει κοινή συμβιβαστική τροπολογία που ε, τη συμπλήρωσαν οι σοσιαλδημοκράτες για, τις, ε, για τα στοιχεία των συναλλαγών, υποβολή λεπτομερών στοιχείων συναλλαγών. Τώρα αν πρέπει αυτά τα στοιχεία να μεταβιβάζονται ή όχι, αυτό βεβαίως ε, ανήκει στο, στην νομοθετική πρόταση της Κομισιόν. Και το ερώτημα είναι αν οι άλλες ομάδες το δέχονται θα μπορούσαμε να κάνουμε την εξής, το συμπληρώσουμε ως εξής και να πούμε το νέο κείμενο όπου, α, όπου χρειάζεται η υποβολή των απαραίτητων λεπτομεριακών ε, στοιχείων της ε, συναλλαγής. Μετά έχουμε την συμβαστική 8 που αφορά το εκτιμώντας 1β, είναι, είναι νέα, νέο εκτιμώντας το οποίο το δέχονται όλοι. Μετά έχουμε τις παραγράφους, συμβιβαστική τροπολογία 9, τη δέχονται όλοι και συμπληρώνει τις τροπολογίες 57 μέχρι 83. Στη συμβιβαστική 9 παράγραφος 1 Έχουμε έτοιμα ξεχωριστής ψηφοφορίας. Το πρώτο μέρος το δέχονται όλοι, το υποστηρίζουν όλοι. αλλάζει την παράγραφο 2. Α, συγγνώμη, διορθώνει ο μιλητής, είναι η συμβιβαστική 10, παράγραφος 2. Εδώ προτείνεται ε, και τη δέχονται όλοι το πρώτο τμήμα το δέχονται όλοι και το δεύτερο, η ξεχωριστή ψηφοφορία, γίνεται δηλαδή μετά από αίτημα των φιλελευθέρων και λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα συγκεκριμένο κριτήριο για την εξέλιξη της ρευστότητας. Γι' αυτό ακριβώς ε, ήταν μια επιπλέον επισημία των φιλελεύθερων, γι' αυτό ξεχωριστή ψηφοφορία. Μετά, παράγραφος 4, συμβαστική 11. Ε, αυτή την υποστηρίζουν όλοι, εντάξει. Συμβιβαστική 12. Επίσης ε, την δέχονται όλοι, όλες οι ομάδες. Για την παράγραφο 6. Για την παράγραφο 7... Τροπολογία συμβαστική 13, χωρίς προβλήματα, παράγραφος 8, συμβαστική 14, χωρίς ε, ε, αντίρρηση παράγραφος 9 ε, συμβαστική 15 εδώ προσθέθηκε μία πρόταση από την αρχική διατύπωση Α, ανταποκρίνεται και στην Επιτροπή Ανάπτυξης, τροπολογία 7 και θα, η συμπλήρωση λέει στο μέσο του κειμένου να προσθέσουμε και στα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην δυνατότητα δημιουργίας, το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός συστημικού κινδύνου. Εν συνεχεία έχουμε τη συμβιβαστική 14 για την παράγραφο 8 και πάλι εδώ δεν έχουμε προβλήματα και παράγραφο 9 τη 15 το είπαμε αυτό για την παράγραφο 12 συμβιβαστική 16 Εδώ ζητείται ξεχωριστή ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα και το δεύτερο τμήμα δεν το δέχονται οι σοσιαλδημοκράτες. Το πρώτο τμήμα έγινε δεκτό από όλους, υποστηρίζει την Κομισιόν και λοιπά, τα CCPs ε, να τα αναπτύξει λαμβάνοντας σεβόμενοι τις διατάξεις της ΕΣΜΑ και ότι τα CCPs δεν πρέπει να επηρεαστούν δυσανάλογα από τους παίκτες της αγοράς. Ωραία, αυτό δεκτό. Η δεύτερη, το δεύτερο τμήμα που έγινε δεκτό από το ΕΛΚ συμπληρώνει ότι θα πρέπει να, ε, ε, ε, ε να εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό ήταν και το τρίτο μέρος λέει ότι θα πρέπει να προταθούν μηχανισμοί για την σωστή διαχείριση της διαδικασίας ανάληψης κινδύνου. Θα πρέπει λοιπόν, το ερώτημα είναι αν θα εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο ε, αυτοί όσοι είναι υπεύθυνοι για την ανάλυση και εκτίμηση του κινδύνου. Συμβιβαστική 18, επί της παραγράφου 15 γενικά αποδεκτή. Συμβιβαστική 19 ε, για την παράγραφο 16 γενικά αποδεκτή. Όπως συμβιβαστική 20 για τη 17 και συμβιβαστική 21 για την παράγραφο 18. Και συμβιβαστική 22 αναφέρεται στο εκτιμωντας ένα 1α, επίσης δεκτό, συμβιβαστική 23, είναι ένα νέο εκτιμώντας, ΕΛΚ, ε, εκτός από τους πράσινους, οι άλλες ομάδες ε, δέχτηκαν το, το ζήτημα των τρίτων κρατών, τρίτων χωρών. Και υπάρχει ένα αίτημα προσθήκης από τους σοσιαλδημοκράτες και από μερικούς φιλελεύθερους από ένα τμήμα των φιλελεύθερων ή από ορισμένους συναδέλφους που είναι πλήρη μέλη εδώ ε, πρόκειται για μία μεμονωμένη λέξη και προτείνω τη λέξη αυτή να την ψηφίσουμε με ξεχωριστή ψηφοφορία σας διαβάζω το κείμενο μέχρι αυτή τη λέξη διαπιστώνει ότι όλες τις συναλλαγές με παράγωγα τα οποία αναφέρονται σε τιμές Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρονται σε ευρωπαϊκή επιχείρηση ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ευρωπαϊκό κλπ. κλπ, κλπ. Το υπόλοιπο είναι το ίδιο. Πρόκειται για το δεύτερο και. Α, αντί για και να γραφτεί ή, το διαζευτικό ή. Δηλαδή, παραγωγά τα οποία αναφέρονται σε συγκεκριμένο ε, συνάλλαγμα σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ή σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία συμμετέχουν. Αντί το και το δεύτερο λοιπόν αντικατασταθεί με το διδευτικό ή. Ε, συμφωνώ με αυτή την προσθήκη, με αυτή την αλλαγή μάλλον, διότι έτσι πιστεύω ότι θα καλύψουμε ευρύτερο πεδίο. Αυτές είναι οι συμβιβαστικέ τροπολογίες τις οποίες επεξεργαστήκαμε και τι τις συζητήσαμε ενδελεχώς. Με, εάν δεχτείτε αυτές τις συμβαστικές θα τελειώσουμε την ψηφοφορία σε 15 λεπτά. Έχω ολόκληρο κατάλογο εδώ, αλλά παρακαλώ εσείς θέλετε το λόγο, ναι. Ναι, ευχαριστώ. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε και για την ε, διαθεσιμότητά του, την ευχαριστήσω τη Γραμματεία της Επιτροπής και της ομάδας μου τη Γραμματεία για την πολύτιμή τους συνεργασία. Να πω αμέσως ότι από την άποψη της διαδικασίας συμφωνώ με τα όσα είπε μόλις ο κύριος Λάγκε όσον αφορά την δυνατότητα να επαληθεύσουμε την ενσωμάτωση των τελευταίων τροπολογιών που υποβλήθηκαν στην ε, συμβιβαστική δουλειά που έχει γίνει. Με αυτή την άποψη πιστεύω πως η δυνατότητα εξέβρεσης ε, ενό πιο προηγμένου σημείου ισορροπίας για να μπορέσουμε να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια οδηγία η οποία να είναι στο ύψος των προβλημάτων και της σοβαρότητας του, της στιγμής είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω πως αυτή η διαθεσιμότητα της, του εισηγητή μας δίνει ένα περαιτέρω χώρο ε, για κοινή εργασία, για συνεργασία, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία αυτής της έκθεσης έχει αυξηθεί σε σχέση με τη στιγμή όπου ξεκίνησε η δουλειά αυτή. Πιστεύω πως το μήνυμα αυτό το σαφές ήδη έχει σε μεγάλο βαθμό εσωματωθεί στις περισσότερες τροπολογίες. Παραμένουν κάποιες διαφορές ανάμεσα στις ομάδες όπως είναι λογικό. Ορισμένες ε, διαφορές στα μείνουν και μέχρι τέλους, αλλά τώρα είναι σημαντικό η Επιτροπή να καταφέρει να δώσει σαφές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπογραμμίζοντας τα πιο σημαντικά σημεία για την αυριανή ψηφοφορία και θεωρώ πως είναι θετικό ότι ένα μεγάλο τμήμα των τροπολογιών που έχει υποβάλει η ομάδα μου έγινε δεκτό από της, ε, στο πλαίσιο των συμβιβαστικών τροπολογιών που μόλις πριν λίγο μας εξέθεσε ο κύριος Λάγκεν. Ελπίζω ωστόσο ότι θα, αυτές τις τελευταίες ώρες θα υπάρξει χώρος για περαιτέρω συνεργασία. Πρόεδρος. Εγώ είμαι η επόμενη, μια που είμαι σκιώδης από τους φιλελεύθερους. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή και να πω ότι οι σεβαστικές τροπολογίες μπορεί να μην είναι τέλειες, αλλά ήθελα τουλάχιστον να υπάρχει μια καλή συμφωνία. Όμως θέλησε άλλες πέντε τροπολογίες να πάρει από τους ε, σοσιαλιστές και να συμπεριλάβει πράγματα τα οποία είχαν αποφασίσει να μην μπουν την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε έτσι χάνει μια ομάδα. Έτσι χάνεται μια ομάδα από το συμβασμό σας. Ε, υπάρχουν τρεις ομάδες τις οποίες δεν ρωτήσατε γι' αυτό. Και σίγουρα κάποιες από αυτές τις τροπολογίες δεν με ικανοποιούν. Μπορεί να υπάρξουν εναλλακτικέ λύσεις, αλλά πρέπει να κάνετε παραπάνω δουλειά για να μπορέσετε τελικά να βρείτε ποιο συμφωνεί μαζί σας και ποιος όχι. Οπότε τώρα είμαι σε δύσκολη θέση. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει ευρεία συνένεση. Αυτή η συνένεση δυστυχώς αρχίζει να καταστρέφεται. Και μια που είμαι και πρόεδρος εδώ, πρέπει να σας πω από τη θέση της Προέδρου ότι δεν είμαι καθόλου ευτυχής να ψηφίσουμε αύριο κάτι το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχετε όλες τις πολιτικές ομάδες. Όχι, δεν λέω ότι θα το εμποδίσω. Απλώς λέω ότι κάνετε τα πράγματα πιο δύσκολα για τις πολιτικές ομάδες. Και λέω ότι θα έπρεπε να κάνετε παραπάνω δουλειά για να μπορείτε να πείτε ότι έχετε ευρεία συνένεση όπως θέλετε. Λοιπόν, τι πράγματα ήθελα να σας πω. Εντάξει, είπαμε, δεν είναι τέλεια, θα μπορούσα όμως να συμφωνήσω με αρκετούς συμβιβασμούς όπου αναφέρεται το θέμα της ιδιοκτησίας, για παράδειγμα. Ποιανού είναι ένα CCP και πού υπάρχει πρόβλημα συμφερόντων. με τους χρήστες για παράδειγμα ή με ανταλλαγές για τα CCP. Οπότε το θέμα αυτό της ιδιοκτησίας πρέπει να το δείτε ολόκληρο για να ξέρετε κατά πόσο μπορείτε να βάλετε κάποια όρια για τους 20 ψηφισμού ή να δείτε κατά πόσο πρόκειται για χρήστες ή για ανταλλαγές και κατά πόσο αυτοί ε, μπορούν να κάνουν κάτι για να βοηθήσουν. Και ότι πρόκειται στο κάτω-κάτω για το κεφάλαιό τους, πρόκειται για πελάτες ή πρόκειται για άλλους. Οπότε η διατύπωση εδώ πιστεύω ότι δεν είναι τέλεια και όσο και να την τροποποιήσουμε πάλι δεν θα είναι τέλεια. Πάντως το βέβαιο είναι ότι υπάρχουν αυτές οι διαφορές και πρέπει να βρούμε το σωστό τρόπο να τις αντιμετωπίσουμε. Οπότε το τελικό προϊόν είναι ικανοποιητικό, να είναι ικανοποιητικό όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου. Τώρα για τις άλλες τροπολογίες που έχουν να κάνουν ε, με ε, το ρευστό, εδώ να αποσύρω εγώ, γιατί πάλι πρόκειται εδώ πέρα για θέμα διαχείρισης κινδύνου. Ορισμένοι βέβαια δεν φαίνεται να το έχουν καταλάβει και νομίζουν ότι αν βάλουμε αυτόν τον όρο, αυτό σημαίνει ότι 9% των νότησης δεν μπορούν να συμψηφιστούν. Αλλά δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόθεσή μας ήταν να μην υπάρξει πρόβλημα συμφερόντων για τη ρευστότητα. Μπορεί, αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, να μπορούμε να βάλουμε κάποια πράγματα πιο ξεκάθαρα για να μην υπάρχει συστημικός κίνδυνος. Αλλά ίσως αυτά είναι υπερβολικά λεπτομερή. Πάντως, αντί να το καταψηφίσετε, εγώ προτιμάω να το αποσύρω, γιατί ίσως είναι περίπλοκο. Και στο κάτω-κάτω αυτά που λέει μέσα αυτό το σημείο υπάρχουν και αλλού στη διαχείριση κινδύνου για παράδειγμα. Οπότε αν σας βοηθάει οι συνάδελφοι να το αφήσω, αλλιώς θα το αποσύρω. Αν δεν το καταλαβαίνετε... Και βλέπω ότι και η Επιτροπή κουνάει το κεφάλι της, οπότε μάλλον το έχει καταλάβει αυτό το θέμα της ρευστότητα. Αυτά είχα να πω. Σήμερα το βράδυ μπορώ να προσπαθήσω να λύσουμε τα προβλήματα που παραμένουν ή να κάνω άλλες τροπολογίες. Ελπίζω να μην θέλετε να τα αλλάξετε όλα. Υπάρχουν τρία πράγματα και το ένα είναι ότι μία από τις ομάδες σας έδωσε τα παράγωγα. Εμείς φτάνουμε σε διέξοδο. Εγώ μπορώ να δεχτώ την αρχική πρόταση και όχι τη συμβιβαστική που είναι μια πιο σφιχτή διάταξη. Αν έλεγε ως ελάχιστο, όχι όμως με το διαζευτικό, γιατί αν έχετε έναν από τους τρεις όρους διαζευτικά να, να καλύπτονται, τότε είναι αλλιώς. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος το πρότεινε αυτό ήθελε να είμαστε προστατευτικοί παραπάνω. Πάντως στην αρχή είπατε ότι όλα τα παράγωγα αποκαλύπτουν τι προϋποθέσεις ως ελάχιστο. Δείχνοντα ότι μπορεί να κάνουν κάτι παραπάνω. Πάντως προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσα να έχω διαπραγματεύσεις μαζί σας για να καταλήξουμε σε κάτι περισσότερο αποδεκτό αν ο κόσμος αυτά τα τρία τα βρίσκει υπερβολικά. Αυτά είχα να πω. Στην ομάδα μου το είχαμε τελειώσει, χωρίς βέβαια να έχω δει όλα αυτά τα καινούρια που προσθέσατε εσείς. Λοιπόν, κατάλογος ομιλητών. Η Σκιώδης πρώτα. Παρακαλώ. Okay. Θέλατε να επανέλθετε ή να μπορώ να πάρω το λόγο. Εντάξει. Α, ελεύθερα. Ίσως να έχετε περισσότερα να πείτε στο τέλος. Θέλετε να κάνετε μια σύντομη παρέμβαση. Εντάξει κύριε Λάγκε, μα θέλετε. Ήθελα να σας παρακαλέσω να ψηφίσουμε γιατί δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα στο πλαίσιο της συνένεσης. Έτσι κι αλλιώς. Ένα, ε, το, το, ένα ή το άλλο επίμαχο θέμα πρέπει να το ψηφίσουμε. Είναι σωστό ότι οι σοσιαλδημοκράτες ε, σήμερα το πρωί πρότειναν περαιτέρω προσθήκες, προσπάθησαν να βρω μια λύση, τα υπόλοιπα είναι ξεκάθαρα. Το θέμα είναι πώς θα ψηφίσουμε αυτά τα επίμαχα σημεία. Η, το τελευταίο σημείο ήταν αυτό το και ή. Εάν βρούμε μία διέξοδο η οποία να είναι σεμιτή. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να διαχειριστούμε θεμητά όλα τα αιτήματα, αλλά δεν μπορούμε ή να ψάχνουμε να βρούμε συμβιβαστικές τροπολογίες που να εκνοποιήσουν όλους. Δεν γίνεται αυτό γιατί υπάρχουν διαφορές απόψεων για τους φιλελεύθερους, κυρία Πρόεδρε, έχετε απόλυτα δίκιο. Αφενός το θέμα της ρευστότητας είναι ένα θέμα στο οποίο οι άλλοι δεν είχαν συμμετάσχει, δεν, δεν συμφώνησαν. Αλλά εάν λάβουν την πλειοψηφία δεν το ξέρουμε. Μπορεί μπορεί χωρίς να υπάρχει γενική συμβιβαστική λύση να, τύχουν, να τύχει αυτή η τροπολογία της πλειοψηφίας. Εν συνεχεία, θα ήθελα να ξέρω και η Κομισιόν πώς εκτιμά το θέμα της δευστότητας σαν κριτήριο του συμψηφισμού, του clearing. Αυτό αφενός, αφετερού, ένα άλλο επίμαχο ζήτημα, είναι τέσσερις τροπολογίες ε, των σοσιαλδημοκρατών εάν στην, ε, στο σώμα διαχείρισης ρίσκου θα πρέπει να εκπροσωπούνται ή υποβάλλοντες τα αιτήματα αν πρέπει να συμμετέχουν δηλαδή στο φορέα αυτόν εγώ δέχτηκα ότι θα πρέπει να συμμετέχουν στο φορέα αυτόν οι σοσιαλιστές και έχουν το δικαίωμα θέλω ξεχωριστή ψηφοφορία το ΕΛΚ θα ψηφίσει υπέρ αλλά θέλουμε ένα δεύτερο τμήμα των σοσιαλδημοκρατών να το συμπληρώσουμε το οποίο ε, δεν είναι διόλου επίμαχο και να πούμε ότι επιπλέον θα πρέπει να προταθούν ευλογοί μηχανισμοί για την θεμητή κατανομή της, του κινδύνου. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι μια γενική διατύπωση πάρα πολύ ωραία που μας εκπροσωπεί θαυμάσια τη προσέγγιση του σώματος. Στο, εκτιμό, στο συμβιβαστικό 23 ε, έχουμε ένα αίτημα το οποίο μόλις τώρα είναι φρεσκότατο, μόλις τώρα μας ήρθε αυτό το θέμα του συμπλεκτικού, του και ή του διαζευκτικού ή. Πρέπει να βρούμε μία τελική λύση. Θα πούμε και ή θα πούμε ή. Εάν πούμε και, τώρα θα έχουμε μία διαβάσμιση τριών βασμίδων, ενώ το or, το διεδεκτικό e, θα είναι δύο οι Στο και, δηλαδή αν ισχύσει το και, τότε θα αναφερθούμε μόνο σε ε, ευρωπαϊκά, στην Ευρωζώνη. Όχι ευρώ, λάθος. Α, εννοώ και σε βρετανικές Τερλίνες. Ναι. Λοιπόν, τρεις βασμίδες θα έχουμε ή δύο. Ο συμβιβασμός ήταν τρεις βασμίδες. Οι σοσιαλδημοκράτες προτιμούν τις δύο βασμίδες ρύθμισης. Το ερώτημα είναι, μπορούμε να βρούμε μια λύση μέσω ψηφοφορίας. Πιστεύω ότι θα βρούμε, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Όλα τα άλλα είναι συντακτικές ε, αλλαγές ρευστότητα, προϋποθέσεις για τρίτες χώρες, συμμετοχή στο φορέα των ε, υποβάλλοντες το αίτημα, των υποβάλλοντων αίτημα, των ετούντων ή όχι. Αυτά είναι διαδικαστικά περισσότερο. Αλλά πιστεύω ότι για να έρθουν οι νομοθετικές προτάσεις στο τραπέζι πρέπει να ασκήσουμε κάποια πίεση. Ε, Ευχαριστούμε. Απαντήσατε σε κάποια σχόλια. Τέλο πάντων, έχω και άλλου ομιλητέ τώρα. Τώρα Κέι. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή που βοήθησε τις τελευταίες δέκα μέρες. Έκανε πάρα πολλή δουλειά πραγματικά και είναι κρίμα ότι μέσα σε 24 ώρες έχουν αλλάξει τα πράγματα και έχει ξεγίνει πολύ από την καλή δουλειά που είχε γίνει. Όντως, αν αλλάξουμε το και και το κάνουμε ή διαζευτικό, έχω πρόβλημα. Πρέπει να το ξαναδείτε. Η συζήτηση που έγινε όλη τη βδομάδα κράτησε πολύ. Τώρα να αλλάξει θα ήταν θλιβερό. Υπάρχουν όμως και μερικά άλλα πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο καταλήξαμε στο συμβασμό 18 την προηγούμενη εβδομάδα και ιδιαίτερα μεταξύ των βοηθών και των συμβούλων οι 2.10 με 2.14 τροπολογίες από ό,τι κατάλαβα θα συμπεριλαμβανόντουσαν στην συμβαστική πρόταση 18 ενώ τώρα βλέπω πω όχι οπότε εφόσον η συμβαστική πρόταση αντικαθιστά μέρος του κειμένου δεν καταλαβαίνω τώρα και κάτι άλλο που όμως αν και φαίνεται μικρό μπορεί να έχει μεγάλες συνέπειες όταν μιλούσαμε για την εξαίρεση του τελικού χρήστη εγώ δεν είχα σκεφτεί ότι όλοι οι dealers αγαθών θα συμπεριλαμβάνονταν εκεί. Και αυτοκινητοβιομηχανία και αεροπορικές εταιρείες από ό,τι φαίνεται μπορούν να αποτελέσουν μέρος της συστημικής αγοράς. Οπότε δεν θα έπρεπε να υπάρχει εξαίρεση. Υπάρχουν κάποια θέματα και με την 116 και 117 τροπολογίες που έχουν να κάνουν με ορισμούς. μιλάμε για τα εταιρικά παράγωγα, χωρίς να λέμε τι είναι αυτά τα εταιρικά παράγωγα. Οπότε χωρίς ορισμό πώς νομοθετούμε πάση περιπτώσει νομίζω ότι η προσπάθεια ήταν τεράστια που έγινε για να καταφέρουμε όλοι να συμφωνήσουμε και είχαμε καταλήξει σε ένα καλό συμβιβασμό. Ελπίζω τώρα την τελευταία στιγμή να μην ξεκάνουμε αυτή την τόσο καλή δουλειά που κάναμε. Ευχαριστώ πάντως για την υπομονή του τον εισηγητή. Σκιώδησε, Πασκάλ είναι ο Ευχαριστώ. Όλοι και εγώ ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε. Ήταν πάντα ανοιχτό να συζητήσουμε και να πετύχουμε ευρεία συνένεση. Τώρα, θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό που μας ε, απασχόλησε πολύ για τις τρίτες χώρες. Εγώ είμαι στη μέση. Συμφωνώ και με τις Σάρων Μπόλς βέβαια που λέει ότι αν έχουμε διαζευτικό ή η θέση μας είναι πολύ ανοιχτή. Αν όλες οι ζώνες του κόσμου υιοθετήσουν αυτή τη ρύθμιση υπάρχει ασυμβίβαστο. Θα είχαμε μία πολύ ανοιχτή ευρεία νομοθεσία. Εάν βάλουμε και, αντίθετα γίνεται πολύ στενή η διάταξη. Είναι πολύ δύσκολο τότε να ελέγξει αυτά που θέλει να ελέγξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, ή που θα βρούμε μια συμβαστική λύση ανάμεσα στι δύο αυτέ διατυπώσει που δεν είναι ικανοποιητικέ ούτε μία ούτε άλλη ή δεν θα τα καταφέρουμε και αν δεν τα καταφέρουμε πολιτικά εγώ θα υποστηρίξω και εμεί θα υποστηρίξουμε εκείνη που βοηθά την Ευρωπαϊκή Ένωση να ρυθμίζει όσο γίνεται περισσότερο και θα προτιμήσουμε το διαζευτικό ή. Αλλά είμαστε ανοιχτοί καλύτερα να προσπαθήσουμε να βρούμε μια άλλη διατύπωση που να είναι συμβατή με αυτά που άλλε χώρες, οι ΗΠΑ για παράδειγμα, θα μπορούσαν να υιοθετήσουν. Και έχω και δύο άλλα πραγματάκια. Για τη συμβαστική που συνυπογράψαμε, είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε το θέμα των αγροτικών προϊόντων και των πρώτων υλών. Επιστήνουμε την προσοχή μας επίσης στο γεγονός ότι σε αυτό το κείμενο δεν υπάρχουν γενικές εξαιρέσεις για τους τελικούς ε, χρήστες, αντίθετα με αυτό που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσπαθήσαμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε τις καλές διατυπώσεις για να λάβουμε υπόψη μας την πραγματικότητα και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των τελικών χρηστών για να έχουμε ένα τελικό συμπέρασμα και μια τελική κατάσταση που να λαμβάνει υπόψη όλες τις περιπτώσεις. Έχουμε μια έκθεση λοιπόν που πηγαίνει προς μια μεγάλη τυποποίηση και προσφυγή στο ΣΕΣΕΠ στο... για το συμψηφισμό. Το περιθώριο επίσης ε, τονίζεται περισσότερο από ό,τι κατά το παρελθόν και λέμε ξεκάθαρα ότι η ευθύνη για να επιλεγεί μια αντιστάθμιση όχι για ένα προϊόν είναι θέμα ευθύνης του ΕΣΜΑΣ που θα είναι και ένα βασικό ζήτημα στην επόμενη οδηγία. Είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλλον θα ήταν, αλλά δεν μπορεί. Θα στηρίξουμε λοιπόν την έκθεση στο σύνολό της και αν τώρα για τις τρίτες χώρες θα μπορούσαμε να μην υιοθετήσουμε πολύ περιοριστική θέση που καταστρέφει τελικά το περιεχόμενο και τις ανησυχίες της έκθεσης αλλά να μην εγκρίνουμε και κάτι το οποίο δεν θα μπορούμε να θέσουμε σε εφαρμογή, αν όλοι ψηφίσουν τέτοιο, θα πετυχαίναμε περισσότερη συνοχή στο κείμενό μας και θα είχαμε μια ευρύτερη ακόμα πλειοψηφία. Δεν είμαστε κατά μιας τέτοιας προσπάθειας. Ευχαριστώ. Έχω δύο-τρεις σύντομες παρατηρήσεις. Έχω υποβάλει και λίγες τροπολογίες. Ε, δεν θέλω να παρέμβω σημαντικά, αλλά στην ε, συμβιβαστική 14 θα ήθελα μία καλύτερη διατύπωση. Λέει ότι τα CCPs δεν θα πρέπει, ε, πιστεύω ότι καλύτερα να πούμε, δεν θα πρέπει να ανήκουν στους ιδιοκτήτες. Όπως αυτή τη στιγμή γίνεται στο συμψηφιστικό οίκο ICE στην Αγγλία, η οποία ICE είπε όσον αφορά τους χρήστες, και τους μετόχους θέλει το ποσοστό, το ποσοστό να το κατεβάσει 25% των ιδίων κεφαλαίων. Not be ε, Συμβιβαστική 16, μία γλωσσική ε, αλλαγή μόνο στην πρώτη αλλαγή στο πρώτο τμήμα θα έλεγα should be represented. Θα πρέπει να εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα πρέπει να εκπροσωπούνται και όσον αφορά τη συμβαστική 23 με το, για το νέο εκτιμώντας, αναρωτιέμαι αν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα με το να ζητήσουμε ένα ελάχιστο επίπεδο ε, ε, as a minimum, ως ελάχιστο. Οπότε ε, λύνουμε το πρόβλημα στην κατώτερη βαθμίδα. Ορίζουμε ένα κατώτερο κατόφλι. Και έχω και μία ερώτηση κατανόησης για τον εισηγητή. Στόχος μας είναι να επιτύχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και όσον αφορά τις συναλλαγές τις ε, standard στα παράγωγα το μεγαλύτερο ποσοστό να τα, να τα μεταφέρουμε στις συναλλαγές over the counter, OTC και ε, πιστεύει ότι με αυτές τις προτάσεις θα επιτύχουμε αυτό το στόχο. Ευχαριστώ ο κύριος Σμιτ. Ευχαριστώ ο κύριος Λάγκε έκανε ό,τι μπορούσε. Και, πρέπει να τον ευχαριστήσουμε για αυτή την τεράστια προσπάθεια. Εγώ θα ακολουθήσω τη γραμμή του σκιώδους εισηγητή μου, αλλά έχω ορισμένα προβλήματα με τη διατύπωση του κειμένου με τις συμβαστικές 11 και 20. Εδώ είναι πολύ θαραλέος ο κύριος Λάγκε που λέει ότι το short selling πρέπει να το απογορεύσουμε. Ε, πολύ παράτολμη αυτή η πρόταση γιατί η πρόσφατη ιστορία μας δείχνει την τεράστια ζημιά την οποία, η οποία έγινε. Εμείς τα απαγορεύσαμε αλλά στη Γερμανία μονόπλευρα πρέπει να κάνουμε κάτι για το short selling. Δεν λέω, αλλά ε, ο τόνος, ο τόνος της πρότασης είναι λίγο λαϊκιστικός. Ε, η λέξη speculation, ε, κερδοσκοπία ακούγεται σαν ύβρις. μην ξεχνάμε ότι ορισμένες κερδοσκοπικές ενέργειες που έγιναν στην Ευρώπη ανέτρεψαν την αγορά. Μην ξεχνάτε ότι και η Γερμανία υπήρξε στόχος κερδοσκόπων στη δεκαετία του 90. Εγώ θα σας ακολουθήσω όμως κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Δεν έχω άλλες παρεμβάσεις. Θα επανέλθω στον κύριο Λάγκε. Η Κομισιόν θέλει να πει κάτι. Ο Πάτρικ. Ο κύριος Λάγκε. Πολύ ε, σύντομα. Η συνάδελφος Βίμπερν ζήτησε να μάθει γιατί οι τροπολογίες δεν ελήφθησαν υπόψη δεν ήταν δικό μου θέμα αυτό, η γραμματεία το κανόνισε. Είχαμε την πρόθεση να τη συμπεριλάβουμε ε, στις συμβιβαστικές, αλλά η γραμματεία 108 μέχρι 114 110 μέχρι 114 αποφάσισε να τις, ψηφίσει, να τις ψηφίσουμε ξεχωριστά. Ο κύριος Καφέ είναι σαφές ότι για το και ή το ή οι πράσινοι επειδή υπήρχε το και δεν συμμετείχαν. Γι' αυτό θέλω να το... Γι' αυτό ήρθε και η αντιπρόταση του διαζευκτικού ή. E. Έχουμε λοιπόν τώρα την επιλογή ή θα ψηφίσουμε την συμβιβαστική 23 ως έχει και εν συνεχεία πρόσθετη ψηφοφορία και ή, ή αν θα αλλάξουμε το διαζευκτικό με το, με συμπλεκτικό με το διαζευκτικό και θα ακολουθήσουμε την πλειοψηφία. Ε, αν η πλειοψηφία θέλει το και ή αν η πλειοψηφία θέλει το ή. Και ο κύριος Κλίντς όσον αφορά τις γλωσσικές μεταβλητές η γλωσσική διατύπωση δεν ε, στρεβλώνει το στόχο πιστεύω ότι ο στόχος μας είναι παραμένει απαράλλακτος και μπορούμε να το τονίσουμε αυτό όσον αφορά τους χρήστες. Παρακάτω, στην τροπολογία λέει ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η διακυβέρνηση, ρύθμιση των ιδιοκτητών, ε, πλαίσιο των ιδιοκτητών και δέσμευση της ρύθμισης, δεσμευτική φύση της ρύθμισης. Άρα τα έχουμε ρυθμίσει αυτά. Όμως έχουμε και το παράδειγμα του Αμερικανικού Μητρώου, των CCP, των Clearing Houses, από το 2009 το Μάρτιο, όπου οι έξι μεγαλύτεροι οίκοι δηλώνουν τις συναλλαγές τους και οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες ε, φορείς τα δηλώνουν αυτά ε, στο αμερικανικό πεδίο και το 25% μπορούν να αποτελέσουν κριτήριο για την Κομισιόν. Ο κύριος Κοφέ ζήτησε ότι τουλάχιστον 80% να, ε, να μπουν στο πλαίσιο των CCPs, των Counterparty Clearing Houses. Και η τελευταία παρέμβαση του κυρίου Σμιτ για την κερδοσκοπία, για τη λέξη κερδοσκοπία. Εγώ το είπα αυτό για την Ελλάδα. Εγώ πίστευα ότι εδώ η κερδοσκοπία που έγινε δεν ήταν υπερβολική. Ό,τι γίνεται, έγινε, ό,τι γίνεται, γίνεται. Δεν λέω. Η προσφυγή κατά της Goldman Sachs και του Paulsen στις Ηνωμένε Πολιτείες όπου Γιάννης Κερνά και Γιάννης Πίνη ε, που είναι καθαρά ε, παράνομη κερδοσκοπία δεν λέω αυτή πρέπει να την κατεπολεμήσουμε Εχτες μου είπαν ότι 3,5 εκατομμύρια τόνοι κακάο θα συλλεχθούν στην εσοδεία του 2010 ενώ αυτή τη στιγμή έχουν γίνει παιχνίδια ε, για την εσοδεία του κακάο 70 ε, εκατομμυρίων δολαρίων ε, δισεκατομμυρίων δολαρίων. Συγγνώμη. Ε, αυτή είναι καθαρή κερδοσκοπία. Όταν η αξία της εσοδείας είναι 3,5 και τα παιχνίδια που γίνονται, τα κερδοσκοπικά, ε, ε, είναι 70 δισεκατομμύρια. Τα τρία κρίσιμα σημεία λοιπόν είναι η συμμετοχή στα CCP, η, συμμετοχή, η ρευστότητα και η συμμετοχή στον διοικητικό φορέα των, ε, αυτών που αναλαμβάνουν τον κίνδυνο. Ευχαριστώ. Ίσως θέλει να σχολιάσει τώρα η Κομισιόν για τα όσα αναφέρθηκαν. Να δώσω το λόγο στον κύριο Πέιτερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε πολύ πολύ επικοδομητική συζήτηση, σαφή μηνύματα. Αυτή είναι η σημασία αυτής της έκθεσης και φυσικά η σοβαρότητα του θέματος ε, γίνεται ε, ξεκάθαρη και το τι περιμένει το σώμα εδώ, δηλαδή συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση από τη δική μας πλευρά λοιπόν, είναι όλα ξεκάθαρα. Κάποια σχόλια. Με ευχαρίστηση παρατηρώ ότι είναι πολύ κοντινή η σχέση για την αντιμετώπιση των ομίλων. Ε, των εταιριών. Είχαμε μια συζήτηση πριν από μερικούς μήνες εδώ στο Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό να βρεθεί μια λογική και λειτουργική ε, λύση που δεν θα εμποδίζει τις επιχειρήσεις της Ευρώπης. Εμείς αυτό το έχουμε σεβαστεί και πρόσφατο ο Επίτροπός μου τόνισε πως η προσέγγιση μας είναι πολύ κοντινή, πολύ παρόμοια με αυτή που ακολουθείτε εδώ στην έκθεση. Επίσης είναι πολύ ικανοποιητικό ότι η εξαίρεση των χρηστών των εταιρικών είναι πολύ σημαντική γιατί είναι πολύ σημαντικό να καλύψουμε, να μπορέσουμε να ε, καλύψουμε αυτούς που είναι συστημικοί χρήστες και να χρησιμοποιήσουμε, τη, να, δούμε και επίσης ποιοι το χρησιμοποιούν αυτό ως παραθυράκι και φυσικά δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει το ίδιο λάθος που προκάλεσε την ίδια την προηγούμενη κρίση. Αν δεν κλείσουμε αυτό το παραθυράκι θα, θα δημιουργήσουμε στην ουσία κίνητρο για τη δημιουργία ενός άλλου σκεώδους χρηματοπιστωτικού διαφορετικού συστήματος, μιας άλλης φούσκας. Ε, ε, Τώρα για την ιδιοκτησία ενός, ενός συμψηφιστικού οίκου. Εδώ θα πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά, να δούμε ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο. Είναι μια ε, ε, ηθελημένη αναντιστοιχεία που μπορεί να δημιουργηθεί μέσα σε έναν ε, τέτοιον οίκο. Μπορούμε να δεχτούμε διάφορες ε, λύσεις. Η πρώτη είναι ένα όριο, ανώτατο όριο ιδιοκτησίας. Εδώ υπάρχουν διάφορα νομικά ζητήματα τα οποία εξετάζουμε μέσα στην Κομισιόν. Η ιδιοκτησία των CCP ήδη ισχύει. Ορισμένα χρηματιστήρια ήδη έχουν στην ιδιοκτησία τους τους συμψηφιστικούς οίκους. Τι κάνουμε λοιπόν, τα αποσυνδέουμε αυτά τα χρηματιστήρια, τα αναγκάζουμε να αναθέσουν σε εξωτερικού συνεργάτε τα CCP τους. υπάρχουν πολλοί νομικά ζητήματα που πρέπει να εξετάσουμε εδώ. Ένα άλλο θέμα που πρέπει επίση να εξετάσουμε είναι υπάρχουν αρκετά στεναρέ απαιτήσει διακυβέρνηση με, με τον ίδιο στόχο και αυτό θα πρέπει φυσικά να το εξετάσουμε για το πώ θα τα θέσουμε όλα αυτά σε εφαρμογή. Το να διαλύσουμε τι υφιστάμενες ομίλου δημιουργεί πολύ σοβαρά νομικά και οικονομικά ζητήματα για αποζημίωση δηλαδή στον τομέα των υποδομών αυτών. Θα πρέπει αυτό περαιτέρω να το συζητήσουμε. Άλλο θέμα είναι η ρευστότητα. Κυρία Πρόεδρε, μπορούμε να συμφωνήσουμε στο ότι αν δεν υπάρχει ρευστότητα κανένα ε, συμψηφιστικό οίκο δεν μπορεί να κάνει καθάριση σε ένα συμβόλαιο παραγώγων γιατί δεν έχει τίτλου για να μετρήσει το κίνδυνο. Εφόσον λοιπόν ένα συμψηφιστικό οίκο δεν μπορεί να μετρήσει τον κίνδυνο, δεν μπορεί και να υπολογίσει τα περιθώρια. Αν δεν μπορεί να, να υπολογίσει τα περιθώρια, δεν μπορεί να εκαθαρίσει ένα προϊόν, γιατί έτσι δημιουργείται ένα σημαντικό συστημικό κίνδυνο. Επ' αυτού δεν υπάρχει διαφωνία. Τρίτη παρατήρηση είναι ότι πιθανότατα θα πρέπει να εργαστούμε σε σχέση με τις απαιτήσει τοποθέτηση των οίκων. Εμεί θα θέλαμε περαιτέρω να συζητήσουμε στη διάρκεια της νομοθετικής αυτής διαδικασία τα εξή. Όχι μόνο τη λέξη και η «ή», δηλαδή στενότερος ή ευρύτερος ορισμός, αλλά είναι και το θέμα τοποθεσία, location, και αυτό θα το συζητήσουμε με το σώμα καθώς θα προετοιμάσουμε την πρότασή μας και λαμβάνουμε υπόψη την άποψη του κ. Λάγκη και την, αυτή που περιλαμβάνεται εδώ σε αυτή την έκθεση. Και θα το συζητήσουμε στο γραφείο του Επιτρόπου. Τέταρτη παρατήρηση αφορά το θέμα του CDS. Εμείς ε, από τα μέσα Νοεμβρίου του περασμένου έτους είδα, κοιτάξαμε ποιοι έλαβαν ποιες θέσεις με ποιους και ποιοι ήταν οι αριθμοί που εμπλέκονταν εδώ. Είμαστε στο τέλος αυτής της έρευνας. για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε στο νομοθετικό γήπεδο για να μπορέσουμε, αν πρέπει μάλλον να απαγορέψουμε ή να επιτρέψουμε τη συνέχιση των CDS. Τέλος, ποιοι θα πρέπει να είναι στις επιτροπές κινδύνου. Όχι μόνο η συμπισπισμό, όχι μόνο αυτή, αλλά αν υπάρχει κίνδυνος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και να συμμετέχουν και οι πελάτες των συμφιστικών οίκων γιατί έχουν άμεσα ε, συμφέροντα. Και το έβρος των αποφάσεων που λαμβάνονται εκεί είναι μεγάλο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Τώρα παραδοσιακά ο εισηγητής θα έπρεπε να έχει το τελευταίο λόγο, τελευταία λέξη αν θέλει. Ευχαριστώ. στα, CDS, στα Credit Default Swaps. Η πρόταση είναι του Επιτρόπου Μπαρνιέ και θα παρουσιαστεί το Μάρτιο, οπότε πρέπει να περιμένουμε. Σα θέλαμε λοιπόν να μας υποβάλλετε τα απορίσματα της έρευνάς σας όσο το δυνατόν νωρίτερα για να μπορούμε να αποφασίσουμε. Και ε, κάτι άλλο, το τελευταίο, ο κύριος Πίρσον είναι υπέρ της τροπολογίας της κυρίας Μπολ στη συμβαστική 10 για τη ρευστότητα. Και ότι αυτό θα πρέπει να είναι το πιο βασικό κριτήριο. Θα πρέπει οι ομάδες να, μελετήσουν, να μπορούν να ακολουθήσουν την πρόταση της κυρίας Μπολς για να ε, κερδίσουμε την πλειοψηφία. Κατά στα υπόλοιπα συμφωνούμε. Ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε αύριο, πιστεύω ότι το ξέρετε όλοι και θα παρουσιαστεί στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Θα μπορούσα ε, να